No, no, no, I'm here uh, for uh, interest. Not uh, involved. Okay, colleagues, if I could ask you to take your seats. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα αρχίσω με τις ανακοινώσεις για τη συνεδρίαση των συντονιστών το πρωί. Πρώτον, για τον ορισμό εισηγητών και εισηγητριών αποφασίσαμε δύο γνωμοδοτήσεις να κάνουμε. Μία για την οδηγία για τα, τις δέσμες ταξιδίων, package travel δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 49 δηλαδή ενισχυμένη πλειοψηφία με την ΙΜΚΟ και οι σοσιαλιστές θα το αναλάβουν. Δεύτερο θέμα, κανονισμός που τροποποιεί τον προηγούμενο για τη νέα γενεά ελεγκτών εναερίας κυκλοφορίας ή διαχείρισης των εναερίων συγκοινωνιών. Ε, το ΕΛΚ θα τον ανάβει. και αποφασίσαμε να μην συγγράψουμε τίποτε για τα υπόλοιπα. για το καθεστώς παρατηρητού της στην ΙΚΑΟ για το Ταϊβάν μετά την αίτηση για αυτό το καθεστώς που έκανε το Ταϊβάν το δέχτηκε και η ΚΑΟ. Είπαμε να σταλούν προτάσεις για νέες δραστηριότητες μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου στο Προεδρείο. Οι συντονιστές αποφάσισαν να να στείλουν, να δεχτούν ορισμένους προσκεκλημένους από το UIC για την ευρωβινιέτα ή ευρώσιμο ή ευρωχαρτώσιμο. Είπαμε το Νοέμβριο να συζητηθεί. Γιατί μερικοί ανησυχούσαν ότι επρόκειτο απλώς για μια ανακοίνωση της Κομισιόν και όχι κάτι ουσιαστικότερο. Θα ζητήσουμε λοιπόν αποσαφηνήσεις. Για την επιτροπολογία οι συντονιστές σημείωσαν το σημείωμα υπαριθμών 17 και για το συντονισμό των πτήσεων είπαν ότι θα εγκρίνουμε την πρόταση απόρριψης που κατέθεσαν δύο ομάδες τροπολογίες μέχρι το 19 Σεπτεμβρίου τις 12 το μεσημέρι στα αγγλικά γιατί δεν υπάρχει χρόνος για μεταφράσεις. Και η Κομισιόν θα πρέπει να μας γράψει επεξηγηματικό σημείωμα. Και το Κοινοβούλιο θα τηρηθεί ενήμερο. Ήδη τα είπαμε προφορικά στην Κομισιόν αυτά, θα τα πούμε και γραπτά. Η απόφαση πάντως θα ληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου για το FTL. Στα δε διάφορα των συντονιστών συζητήσαμε και τις απεργίες στις ποτάμιες συγκοινωνίες της Γερμανίας και αποφασίσαμε να μην κάνουμε τίποτα αν όμως οι ομάδες θέλουν να αναλάβουν καμιά πρωτοβουλία ας την αναλάβουν. Αυτά για τους συντονιστές. Φαντάζομαι γίνονται δεκτά και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η παρουσίαση μελέτης του θεματικού τμήματος για τα οχήματα μεγάλου μήκους. Μπορεί να θυμάστε ότι είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η μελέτη λόγω της αβεβαιότητας ή και των αντιμαχωμένων απόψεων που είχαν ακουστεί για το θέμα των μεγάλου μήκους φορτηγών που κυκλοφορούν διαμεθοριακά πέρα από όσα προβλέπει η σχετική οδηγία. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και η Κομισιόν πρότεινε αλλαγή στο βάρος και διαστάσεις των οχημάτων αυτών πράγμα που μας δίνει και την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Επομένως αμέσως τώρα οι συντάκτες της μελέτης θα την παρουσιάσουν. Το πολύ για 15 λεπτά. Θα είμαι αυστηρότατος με το χρόνο. Γιατί συνήθως έρχονται άνθρωποι να μας παρουσιάσουν απόψεις και μελέτες και είτε τους έχει δοθεί περιορισμένος χρόνος είτε όχι το ίδιο τους κάνει. Θα τα πούν όλα. Όχι, 15 λεπτά για τον Steve Davis. Μετά τέσσερις άλλοι, όχι, συγγνώμη. Μετά ο εισηγητής για πέντε λεπτά και μετά οι άλλοι. So, um, who's doing it for Steve Davis? Μετά οι reviewers now. Για να πούμε και για τους επισκέπτες. Έχουμε εδώ επισκέπτες της κυρίας Βανόη που κάλεσε 23 τοπικούς ελεγκτές των γαλλικών σιδηροδρόμων. Πολύ αστείο που είστε από τους σιδηροδρόμους ενώ εμείς θα μιλήσουμε για φορτηγά, αλλά τέλος πάντων. Ντέιβις. The projected. There you go. Να και οι διαφάνειες. Καλησπέρα σας. Ε, ονομάζομαι James Steers από την Steer Davis Cliff και θα σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας για τον αντίκτυπο των μεγάλων φορτηγών. Θα δείτε ποια είναι, ποιος είναι ο μορφότυπος της παρουσίασης. Θα σας δώσω λοιπόν και κάποια αποτελέσματα, τα αποτελεκτικά στοιχεία τα οποία βρήκαμε σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των μεγάλων αυτών οχημάτων, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Και μετά θα κοιτάξω ποια είναι η σχέση μεταξύ των μεγάλων αυτών φορτηγών και τη ε, πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με αυτά θα κλείσω. Οχτώ Έχουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά ε, και μια ισορροπία για την μελέτη. Κοιτάξαμε λοιπόν μελέτες με μεγάλο εύρος ε, αντικειμένου και ε, με διαφορετική γεωγραφική κάλυψη. Στην Ευρώπη, στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες και κάποιες είχαν και ένα πεδίο εφαρμογή παγκόσμιο. Επίσης, λάβουμε υπόψη και υπέρ και κατά των φορτηγών μελέτες. Όλες οι μελέτες που εξετάσαμε υποδεικνύουν ότι οι χρήσει ε, φορτηγών θα αύξαν το κόστος ένα χιλιόμετρο επειδή απαιτείται πιο μεγάλη μετακίνηση μεγαλύτερων φορτηγών και πιο πολύ καύσιμο κατά συνέπεια. Ωστόσο θα έπεσε το κόστος ανά χιλιόμετρο τόνου γιατί ε, τα μεγάλα αυτά οχήματα περιλαμβάνουν τριπλό όγκο σε σχέση με τα κανονικά φορτηγά. Ωστόσο δεν κοστίζουν κατά 50% λιγότερο σε σχέση με τα λιγότερα με τα κανονικά φορτηγά. Και όλοι συμφωνούν ναι, ο πρόεδρος ε, υποδεικνύει ότι σας είπα ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε σε 15 λεπτά, αλλά σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά. Όλες οι μελέτες επίσης συμφωνούν ότι η εισαγωγή μεγάλων φορτηγών θα οδηγήσει σε κάποια μετατόπιση από τις μεταφορές της εναέριες και τις τηλεδρομικές στις οδικές μεταφορές. Ωστόσο, παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη διαφωνία για το ποσοστό της μεταφοράς αυτής στις οδικές μεταφορές. Τέλος, οι μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν μεγάλα κενά σε ό,τι αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα μεγάλα αυτά φορτηγά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι βασιζόμαστε σε μελέτες ενημερωτικές, αλλά που δεν μπορούν να προβλέψουν το πραγματικό αντίκτυπο της χρήσης των φορτηγών. Ο συνολικό όγκος των μεταφορών είναι λίγο πολύ ο ίδιος τα τελευταία χρόνια με μία μικρή μείωση λόγω της οικονομικής κατάστασης. Το 2007 φτάσαμε στο άνωτατο επίπεδο και το 73% λοιπόν ε, γίνεται, των μεταφορών γίνεται μέσω των ε, φορτηγών, 6% μέσω του νερού και πρέπει να σας πω ότι συνολικά οι έξι μεγαλύτερε αγορέ ε, για τις οδικέ μεταφορέ είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Πολωνία. Καλύπτουν το 80% των συνολικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μόνο η Γερμανία επιτρέπει τη χρήση των μεγάλων φορτηγών και πάλι όμως σε περιορισμένη βάση. Δοκιμαστική. Και επιτρέπονται μόνο στη Φιλανδία και στη Σουηδία. Ανά χιλιόμετρο τόνο αντιστοιχούν σε 73% στη Σουηδία. Το ποσοστό αυτό είναι πιο υψηλό. Τα μεγάλα φορτηγά έχουν μερίδιο της αγοράς 90% σε τόνο χιλιόμετρα. Τα φορτηγά και τα μεγάλα φορτηγά χρησιμοποιούνται λοιπόν στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Δανία. Το 2008 ξεκίνησε στην Ολλανδία να δοκιμάζονται και μέχρι το 2010 ήταν 3,6% και 450 ήταν τα μεγάλα αυτά φορτηγά στους ε, δρόμους της Δανίας. Το, στις αρχές του 2013 ήταν 600 στον αριθμό. Οι, γερμανικές, δοκιμές ξεκίνησαν στις αρχές του 2012 και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτος στη Γερμανία είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός, 38. Άρα και ο συνολικός όγκος μεταφοράς είναι περιορισμένος. Ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε το 2001 τέτοιες δοκιμές με τέσσερα συμμετέχουσες εταιρείε. Και μετά ήταν πιο μεγάλη η συμμετοχή και το 2007 ξεκίνησε μια νέα περίοδο δοκιμής. Τον ε, Ιανουάριο του 2010 είχαμε 196 τέτοιες εταιρείε και πάνω από 400 τέτοια φορτηγά σε όλη την, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα εξή στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση, για παράδειγμα, μεγαλύτερων τρένων σημαίνει χαμηλότερο κόστος από τη χρήση τέτοιων φορτηγών. Αλλά σημαίνει ότι αυτό προαπαιτεί κάποια συγκεκριμένη συχνότητα για τα τρένα αυτά. Αν περιορίζονται λοιπόν τα μεγάλα αυτά φορτηγά στους ε, δρόμους, θα έχουν μικρότερο δυναμικό ε, εισχώρηση στην αγορά. Τα μεγάλα φορτηγά έχουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κανονικά φορτηγά σε ό,τι αφορά μεγάλα ταξίδια και ό,τι αφορά προϊόντα μικρής πυκνότητας, γιατί αυτά χρειάζονται μεγαλύτερο τον επιπλέον όγκο που προσφέρουν τα μεγάλα φορτηγά και τα στοιχεία της Φιλανδίας υποδεικνύουν ότι κυρίως στην γεωργία, στα τρόφιμα και στα κλωστοφαντουργικά προϊόντα χρησιμοποιούνται αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Πώς μεταφέρονται τώρα τα φορτία στην Ευρώπη. Η κατανομή είναι λίγο πολύ ίδια τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα τρία τη μεγαλύτερη ποσοστό σιδηροδρομικών μεταφορών είναι η Λιθουανία, η Λεκτονία και η Εστονία. Και γενικά τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης προτιμούν τους σιδηροδρόμους ενώ αυτό το ποσοστό είναι πιο χαμηλό στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σουηδία και η Φιλανδία έχουν 35-25% σιδηροδρομικών μεταφορών παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν και τα μεγάλα αυτά φορτηγά και φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές στο ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στους τρόπους μεταφοράς. Αυτό εξαρτάται και από τη ζήτηση για τη μεταφορά τέτοιων φορτίων. Δύο παράγοντες είναι σημαντικοί για τον αντίκτυπο των μεγάλων αυτοφορτηγών. Το κόστος σε σχέση με όλες τις ε, τρόπους μεταφορών. Καταρχάς λοιπόν έχουμε ε, το πόσο η τιμή θα αλλάξει τη ζήτηση. Ενώ ο άλλος παράγοντας έχει να κάνει με το πόσο η αλλαγή στην τιμή των ειδικών μεταφορών θα αλλάξει τη ζήτηση για τις ειδομικές μεταφορές. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, πολύ περιορισμένε ε, τέτοια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, αλλαγή της ζήτηση. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν συμφωνούν όμως οι έρευνες σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των μεγάλων φορτηγών και αυτό λοιπόν σημαίνει μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για την αλλαγή στον τρόπο μεταφορά μεταφράσει. Προβλέπεται σε κάποιες περιπτώσεις 20-30% μείωση των συνδρομικών μεταφορών, 20-30% θαλάσσιων μεταφορών, 10-15% στις μεταφορές τροφίμων και 10-15% στα τρόφιμα χήμα. Αυτό το προέβλεψε η CEA, ωστόσο. Αντιθέτως, το, Ευρωπαϊκό, το Ολλανδικό Υπουργείο Μεταφορών Κατέλήξε στο συμπέρασμα ότι το 90% των μεταφορών δεν θα ε, επηρεαζόταν από τα μεγάλα αυτά φορτηγά. Παρακολουθούμε όμως τον αντίκτυπο αυτό. Η σουδική τώρα εμπειρία. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν απαγορευτούν τα μεγάλα φωτοφορτηγά από τους ειδικούς δρόμους, δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά ιδιαίτερα το σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί οι σιδηρόδρομοι ήδη λειτουργούν στην, ε, στο πλήρε των δυναμικών. Και άρα καταλήγουμε στο ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε μόνο τον αντικτύπο των μεγάλων φορτηγών, πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και με τους άλλους τρόπους ε, μεταφορών. Και έτσι ενδεχομένω να είναι μικρός ο αντικτύπος σε περίπτωση εισαγωγή των μεγάλων αυτών φορτηγών. Ή ενδεχομένω να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ζήτηση για μεταφορές. Και αυτό ε, εξαρτάται από την ελαστικότητα της ε, ζήτησης. Και σε αυτό πραγματικά δεν καταλήγουν σε κάποια ενιαία τοποθέτηση οι μελέτες. Τώρα, το εξωτερικό κόστος των μεταφορών είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική πτυχή, αν θέλετε, για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Καταρχάς, κοιτάξουμε το κόστος σε ό,τι αφορά τις υποδομές, το κόστος σε ό,τι αφορά στις αλλαγές της ροής των ε, δρόμων μετά από την εισαγωγή των μεγάλων φορτηγών, το κόστος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους δρόμους και το κόστος που συνδέεται με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Σε ό,τι αφορά τις υποδομέ έχουμε τρεις τομείς. Μακροπρόθεσμα, στους δρόμους, στο χώρο και στον ε, στις πλατείες και το καταξής ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε πάρκινγκ, σε τέρμιναλ και ο αντίκτυπος σε δομές όπως για παράδειγμα οι γέφυρες που θα πρέπει να βελτιωθούν. Ο βαθμός στον οποίο θα γίνει μεταφορά προς αυτόν τον τρόπο μεταφορών, ε, μετάβαση προς αυτόν τον τρόπο μεταφορών, θα έχει να κάνει και με το κόστος. Και τα χαρακτηριστικά φυσικά των μεγάλων φορτηγών μπορεί να επηρεαστούν και επειδή φυσικά είναι πιο βαριά αυτά τα οχήματα. Άλλες έρευνες ε, θεωρούν ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και άλλες όχι. Σε ό,τι αφορά και τη χρήση των αξώνων που θα είναι 7 και όχι 4. Ε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι μικρότερη επιβάρυνση ανά άξονα σε σχέση με τα παραδοσιακά φορτηγά. Τώρα τι γίνεται με τις γέφυρες, με τα τούνελ, μπορεί να αντέξουν το επιπλέον βάρος. Αυτό μπορούμε να το περιορίσουμε και περιορίσοντας το δίκτυο που μπορούν να ε, κυκλοφορήσουν τα φορτικά αυτά. Για να αποκλειστούν, για παράδειγμα, οι γέφυρες και τα τούνελ. Τι γίνεται με τους χώρους στάθμευσης. Αυτό διαφέρει πάρα πολύ αναχώρα. Όπως, ε, χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα που έχουν μεγάλες ορεινές περιοχές, πολλά τούνελ, θα αναγκαστούν να περιορίσουν σημαντικά και να αλλάξουν σημαντικά το δεκτύο τους. Τώρα, τι γίνεται με τις ε, ροές κυκλοφορίας. Κοιτάμε τις μελέτες και διαπιστώνουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο, για παράδειγμα, να προσπεράσουμε τέτοια φορτηγά. Αλλά δεν φαίνεται αυτός ο δίκτυπος να είναι σημαντικός. Τώρα, τι γίνεται με τα ατυχήματα, με την ασφάλεια στο δρόμο. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα τα φορτηγά αυτά. Παρ' όλα αυτά, δεν βρήκαμε στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι θα είναι σημαντικά, θα επηρεαστεί η ασφάλεια στους δρόμους μετά από την εισαγωγή των φορτηγών αυτών. Ούτε στη Σουηδία, ούτε στη Φιλανδία φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και πιο πολλά περιστατικά. Τα πιο πολλά ποσοστά θνησιμότητας ε, μοιραίων ατυχημάτων θα προκαλούνταν και από κανονικά φορτηγά και οι πιο πολλέ μελέτε κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φορτηγών αυτών ενδεχομένως να βελτιώσει και την ασφάλεια επειδή θα είναι πιο λίγα στον αριθμό τα φορτηγά που θα κυκλοφορούν. Ο αντίκτυπος τώρα σε ό,τι αφορά την εκπομπή ε, αερίων του θερμοκηπίου εξαρτάται από τρεις τομείς. Η μείωση ε, των ε, καυσίμων ανά χιλιόμετρο, ε, η διάδοση των ε, αερίων αυτών και η αύξηση λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης για μεταφορά φορτίων. Και οι μελέτες καταλήγουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. μελέτες ε, κατέληξαν σε συμπεράσματα από 0,5 έως 1,5 έως και 4% σε ό,τι αφορά την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Οι οδικές μεταφορές ε, είναι υπεύθυνες για μεγάλο τμήμα των εκπομπών αυτών και έτσι η αύξηση που θα προκληθεί από τη χρήση μεγάλων φορτηγών θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική εκπομπή και σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι προβλέπεται αύξηση από 0,4% έως και μείωση μείων 1,2%. Άρα σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή η χρήση των φορτηγών αυτών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσον βοηθούν και θα συνδράμουν στην επιτεύξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το αντίθετο να πούμε ότι μάλλον πιο πιθανό είναι να βελτιώσουν την κατάσταση. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους δρόμους. Κλείνοντας, οι απόψεις πραγματικά είναι διστάμενες σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, τα πορίσματα των μελετών. Και το βασικό είναι το τι θα γίνει και με όλα τα, τους παράγοντες ελαστικότητας. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πιο στενά τις ε, μελέτες που γίνονται στην Ολλανδία και στην Δανία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ε, uh, ευχαριστούμε πολύ. Ο Like Friday. Πέντε λεπτά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω. Μάλλον συνήθω μιλάω αγγλικά ή προσπαθώ τουλάχιστον να μιλάω αγγλικά, αλλά αυτή τη φορά θέλω πραγματικά να γίνω κατανοητό, γι' αυτό θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Ναι, ε, εννοείται, παρόλο που πολλοί προτιμάνε να μην παρακολουθούν από τη διερμηνία, αλλά εγώ κάθε άλλο παρά θα σας πω να μην μιλήσετε τη μητρική σας γλώσσα. Παρακαλώ. Αλλά προηγουμένως υπάρχουν διάφοροι όρθιοι. Καθίστε στις κενές θέσεις και όταν έρθουν οι ευρωβουλευτές οι κλητήρες θα σας ζητήσουν να σηκωθείτε για να καθίσουν ανάλογα με το που είναι η θέση τους. Οπότε ας το κανονίσουμε λιγάκι, ας βοηθήσουν και οι κλητήρες να καθίσει ο κόσμος. Είναι αστείο να υπάρχουν κενά καθίσματα στην αίθουσα και να είναι τόσοι όρθιοι. Λοιπόν, όταν έρθουν οι προβουλευτές σας καθίσουν από εδώ και στις υπόλοιπες θέσεις να καθίσουν οι επισκέπτες μας. Πέντε λεπτά λοιπόν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν είπα και πρώτη φορά τη μελέτη, σκέφτηκα δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία είναι υπέρ των φορτηγών αυτών και κάποια στοιχεία τα οποία συγκλίνουν μάλλον κατά τη χρήση τέτοιων φορτηγών. Και ήταν καθήκον μου να μην το κοιτάξω μόνο επιφανειακά το θέμα αυτό τη μελέτη, αλλά να επισέλθω στις λεπτομέρειε. Και όταν ξεκίνησα λοιπόν να την εξετάζω, κατέληξα στο εξή συμπέρασμα σε χαρακτήρια. Σε χαρακτήρια σε εκείνους που, τις, ε, που την συνένταξαν γιατί? Γιατί έκαναν κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί ποτέ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία εξαιρετικά εξονοχιστική, αν θέλετε, προετοιμασία μιας τέτοια μελέτης και τελικά μία εξονοχιστική μελέτη. μελέτη. Και γιατί το λέω αυτό? Κοιτάξαμε πώς συντάχθηκε λοιπόν η μελέτη αυτή. όπως και άλλες μελέτες που έχουμε δει. Μαζέψαν κάποιες μελέτες, τις ε, οποίες και τελικά ε, ξεκαθάρισαν, καταλήξαν σε κάποιες συγκεκριμένες, αλλά έχουν θέσει κάποια πολύ καλά κριτήρια. Τρία συγκεκριμένα. Να υπάρχει μια ευρεία παλέτα θεμάτων στην μελέτη αυτή, γεωγραφική ε, πεδίο να είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει και μία διάκριση και να συμπεριληφθούν και οι υπέρμαχοι αλλά και οι πολέμοι των φορτηγών αυτών και επιλέχθησαν κάποιες μελέτες έτσι με τον τρόπο αυτό. Έξι υπέρ, μία εν μέρη υπέρ εν μέρη κατά και μία κατά. Άρα εννοείται όταν ξεκινώ από την επιλογή των μελετών να επιλέγω με έξι υπέρ και μία κατά, προφανώς θα υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τρεις ήταν γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ήταν από την Αυστραλία. Μα πού είναι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέσσερις ρήμους όπως έχουμε στην Αυστραλία. Και τρεις τρία, τρεις μελέτες από Ηνωμένα Βασίλεια, Ολλανδία και Σουηδία, δηλαδή από τις χώρες αυτές που χρησιμοποιούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Μα τι το αντικειμενικό υπάρχει λοιπόν σε, αυτές τις, σε αυτή τη μελέτη. Έχει και ακολουθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εξ αρχής ένα στοχό είχε. Όχι να εκπληρώσει την εντολή του Ευρωπαίου Φορολογούμενου και τη σύνταξη πραγματικά αντικειμενική μελέτη, Από ό,τι φαίνεται, τελικά καταλήξαμε σε μια μελέτη που βοηθάει όλους όσοι θέλουν να προωθήσουν τελικά αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Και γιατί υπάρχουν στοιχεία πριν από το 2010 τα οποία συμπεριληφθήκαν στην μελέτη. Υπάρχουν τόσα καινούργια μεγάλα, πιο, τόσο πολλά πιο πρόσφατα στοιχεία γιατί υπάρχουν και επικριτικά στοιχεία. Ποιος έκανε την επιλογή αυτή και γιατί. Και μόνο τότε μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και πορίσματα και δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρεια αλλά για παράδειγμα το συμπέρασμα ότι στην ε, Ολλανδία η προσαρμογή στις κάτω χώρες, στις υποδομές και στους δρόμους δεν ήταν ιδιαίτερος μεγάλη, είναι μια τρασίτητα. Η Ευρώπη, τι να σας πω, δεν είναι όλοι επίπεδοι, δεν είναι όλοι επίπεδοι και δεν έχει εισάγει το όριο των 50 τόνων πριν από κάποια χρόνια όλοι. Αυτό δεν είναι καν επιστημονικά ορθό. Κοιτώντας επίσης το model shift, την αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς. Αν ε, κάνουμε υπολογισμούς, να ξέρουμε ότι οι σιδηρόδρομοι στην χώρα αυτή δεν ε, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για μεταφορά φορτίων όπως σε άλλες χώρες. Πώς να κάνουμε μια τέτοια υπολογισμό λοιπόν. Μόνο τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει περιορισμό περιορισμένος αντίκτυπος στου σιδηροδρόμους μόνο όταν μιλάμε για χώρες όπου δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό μεταφορών σιδηροδρομικών των φορτίων. Δεν είναι το μέσο αποτέλεσμα αυτό στον οποίο καταλήγουμε. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουμε βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, των συγκεκριμένων χωρών. Σε καμία περίπτωση δεν πήρατε υπόψη στη μελέτη σας αυτά που είναι σημαντικά για μας στοιχεία του πώς θα επηρεαστούν οι εργασιακές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό για τις θέσεις εργασίας, τις θέσεις εργασίας, τους ιδιόδρομους, στην όλη η οικονομία των μεταφορών. Όλα αυτά δεν τα λάβατε υπόψη. Και η δική μου εντύπωση είναι η εξή. Ήταν πραγματικά κακή η μελέτη αυτή υπέρ των λόμπι για των φορτηγών αυτών και δεν βλέπω γιατί θα πρέπει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος να πληρώνει μια τέτοια μελέτη. Thank you. I to... Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στους ε, τέσσερις που για πέντε λεπτά ο καθένας θα σχολιάσουν. Ο καθηγητής Γροζέ πρώτα. Σας ευχαριστώ όλους. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά στη μητρική μου γλώσσα. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Η μελέτη που ξαναδιάβασα ξεκίνησε από μια εντολή η οποία πιστεύω ότι τηρήθηκε αρκετά. Πρώτα απ' όλα προσπαθούσε να απομονώσει τις επιπτώσεις που έχουν τα μεγατράξ αυτά στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στις μεταφορές και προσπάθησε να καταλήξει σε μια πιο μεγάλη, πιο ευρεία άποψη και πρέπει να σας πω ότι εγώ προεδρεύω το παρατηρητήριο στη Γαλλία για τις μεταφορές και μας ζητήθηκαν πριν από τέσσερα χρόνια να κάνουμε ακριβώς την ίδια μελέτη στη Γαλλία. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο όπως στη μελέτη που εξετάζουμε σήμερα. Τεχνικά δηλαδή μιλώντας, αυτά τα μεγάλα φορτηγά δεν δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υποθέτουμε ότι δημιουργούν. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντα οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να μην αυξηθούν σε ορισμένε περιπτώσει και η μεταφορά από το ένα μέσο μεταφορά στο άλλο να μην επηρεαστεί ιδιαίτερα. Η αδυναμία τη μελέτη ίσω να έγκυται στο δεύτερο τμήμα που είναι πιο σύντομο και έχει να κάνει με τα σενάρια. Θα το διαπιστώσατε ότι τα σενάρια λένε ή δεν κάνουμε τίποτα, do nothing, ή ανοίγουμε λίγο την πόρτα ή την ανοίγουμε πάρα πολύ την πόρτα στα φορτηγά αυτά. Τα σενάρια αυτά λοιπόν τι μας λένε. Μας λένε ότι πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, αν τα, τα συσσωρεύσουμε το ένα δίπλα στο άλλο, υπάρχει το πολιτικό ζήτημα, η πολιτική επιλογή. Και εδώ θα είμαι σύντομος. Είναι αποδεκτά τα φορτηγά αυτά να ανοίξουμε την... το κουτί της Πανδώρας για τους σιδηρόδρομους, διότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές μειώνονται στις χώρες μας, έχουμε διαπιστώσει, οπότε μόνο να ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας υπέρ των σιδηροδρόμων. Οπότε, αν τελικά οι μεταφορές δεν πάρουν, οι συνδρομικές μεταφορές δεν πάρουν κομμάτι των μεταφορών, τότε ναι, ίσως πρέπει να πούμε ότι αυτά τα φορτηγά μπορεί να αποτελέσουν κάποια λύση. Πάντως ο οργανισμός του οποίου προεδρεύω εγώ τελικά σύστησε στον Πρωθυπουργό να μην κάνουμε τίποτα. Do nothing. Σήμερα στους δρόμους κυκλοφορούν διαφορετικού είδου χρήστε. Εγώ είμαι οικονομολόγο και πρέπει να σα πω ότι καθαρά οικονομικά μιλώντα, η... τα αποτελέσματα για τον χρήστη είναι τα πιο σημαντικά. Αυτό που έχει σημασία για του πολιτικού, δηλαδή είναι το ποιο ψηφίζει. Ψηφίζουν οι χρήστες, οι πολίτες και δεν ψηφίζουν τα φορτηγά. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα όμως που είναι από πίσω και δεν είναι μόνο αυτό των μεγάλων φορτηγών και είναι αυτό της βελτίωσης του ποιοτικού άλματος που πρέπει να γίνει στην μεταφορά εμπορευμάτων είτε έχουμε τα μεγατράξ είτε δεν τα έχουμε, στον τομέα της ασφάλειας. Αν τα μεγάλα αυτά φορτηγά μπορούν να αποδείξουν ότι οι δρόμοι μας γίνονται πιο ασφαλείς όταν έτσι μεταφέρονται τα εμπορεύματα, γιατί όχι αλλά βλέπετε ότι το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό και τα τεχνικά ζητήματα απλώς δείχνουν τι είναι το εφικτό βήμα-βήμα, ενώ η πολιτική επιλογή είναι τελικά αυτή που βαρύνει. Δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο, με καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Τώρα ο καθηγητής Ότε άλλη Μακίνεν από το Λογιστικό Πανεπιστήμιο Κούν. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά εντυπωσιάστηκα από αυτή την παρουσίαση. Ήταν πολύ δύσκολη η μελέτη λόγω της πολλή δουλειάς που χρειάστηκε και της διαφοράς με τα προηγούμενα δεδομένα. Αλλά η εντολή που δόθηκε τελικά ήταν ανεπαρκή, ανεπαρκής γιατί βασίστηκε στο κόστος των μακρών φορτηγών Εξάλλου και η ορολογία mega track δεν είναι και πολύ αντικειμενική. Είναι συναισθηματική. Δεν ζήτησαν όμως να μελετηθούν και τα οικονομικά ωφέλη των μακρών αυτών οχημάτων. Οι τρόποι δηλαδή με τους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί η οικονομική συνοχή της Ένωσης. Υπήρχε λοιπόν από την αρχή, από την ίδια την εντολή της μελέτης, κάποια στρέβλωση που θα οδηγούσε σε αρνητικά εκ των προτέρων αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά έκαναν ό,τι μπορούσαν και μελέτησαν τις προηγούμενες μελέτες που ήταν οι πιο επιστημονικά αυστηρές. Εκείνες που αποκλείστηκαν νομίζω δικαίω αποκλείστηκαν. Άλλο, ποιος πλήρωσε τις μελέτες, τη μελέτη. Ένα είναι αν ήταν κομισιόν και κυβερνήσεις και άλλο θα ήταν αν τις είχαν χρηματοδοτήσει ομάδες πίεσης και λόμπι. Είναι λοιπόν συνοπτική και περιεκτική η μελέτη, αλλά κατ' εμένα θα ήθελα τα επιχειρήματά της να ενδυναμωθούν. Να σας αναφέρω μερικά. μερικοί μίλησαν για τον οικονομικό αντίκτυπο όχι μόνο τις εξοικονομήσεις στο κόστος αλλά και έμεσα ωφέλη από την αναδιάρθρωση της λειτουργίας των εταιριών. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να το δουν πιο λεπτομερώς. Είναι εκείνες οι αξίες για την ελαστικότητα που μας ανέφεραν. Εδώ υπήρχαν τρομερές διαφορές. Δυστυχώς νομίζω ότι στον τομέα αυτόν βασιστήκαμε υπερβολικά στην οικονομετρία και λιγότερο στα στοιχεία των ίδιων των ενδιαφερόμενων. Πού χρησιμοποιούν και πότε τα οχήματα αυτά οι εταιρείε και γιατί έτσι θα καταλαβαίναμε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Το βάρος τώρα. Και εγώ πριν από μερικά χρόνια ανέλαβα μια σχετική μελέτη και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς ποιο ακριβώς είναι το αντίκτυπο από την λειτουργία αυτών των μακρών φορτηγών. Γιατί υπάρχει και το θέμα της πυκνότητας ή μεγαλύτερης ή μικρότερης πυκνότητας κυκλοφορίας γενικότερα στους δρόμους. Το θέμα βέβαια το έχουν κοιτάξει πολλοί, δεν χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής για να το καταλάβει, αλλά χρειάζονται καινούρια στοιχεία για την πυκνότητα της οδικής κυκλοφορίας. Και στα επόμενα λεπτά που μου απομένουν, θα έλεγα ότι όλα εξαρτώνται από τη σημασία που δίνουμε στον λόγο κόστους ελαστικότητας. Μεγάλο μέρος της ανάλυσης υπέθεσε ότι οι οδικές μεταφορές εξαρτώνται απόλυτα από την τιμή ενώ παραγνώρισε το θέμα της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Σύστημα μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει πολύ ψηλή ποιότητα. Βελτιώνεται όμως, βελτιώνεται αν από την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των μεγάλων φορτηγών μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση για τους σιδηροδρόμους, θα να ελαφρύνουμε. Θα μπορούσαν και αυτοί να βελτιώσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρουν και μερικά γενικά και καταληκτικά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πιο θετικές μελέτες για τα βαρέα φορτηγά είναι εκείνες που βασίζονται σε δείγματα πραγματικά δεν είναι θεωρητικές έννοιες τα βαρέα φορτηγά. Πρέπει να δούμε σε ποιες χώρες την Ένωση αλλά και αλλού για να μην αγνοήσουμε και την εμπειρία χωρών εκτός της Ένωσης. Ποια χώρα απελευθέρωσε πλήρως την τη λειτουργία τους και μετά μετάνιωσε. Καμία νομίζω. Άρα υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι τα οχήματα αυτά πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Και κάτι άλλο. Αντί να συζητάμε για το αν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν ή όχι, πρέπει να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε ένα είδος βαριού φορτηγού το οποίο να είναι πιο αποδοτικό και πιο αποδεκτό. ώστε να λειτουργεί πιο ολοκληρωμένα μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα και επίσης να μειώνει και τις επιπτώσεις που επιβαρύνουν την κατανομή σιδηροδρόμου και όχι αυτοκινήτου. Τώρα ο Τιμ Μπρίμερ από τη Λουβένη. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Γενικά μιλώντας, θα έλεγα ότι βρήκα τη μελέτη αυτή χρήσιμη. Τις επιπτώσεις δηλαδή από την εισαγωγή των Megatrax. Τέθηκαν τα κυριότερα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα από αυτά που διάβασα, συμφωνώ με τον καθηγητή Μακίν, τα ίδια θα έλεγα και εγώ, τους ίδιους περιορισμούς βλέπω και εγώ. Οι επιπτώσεις ποιες είναι. Είναι ότι πολλαπλασιάζεται η κυκλοφορία, είναι το θέμα των επιπτώσεων στην κυκλοφορία αυτή καθεαυτή. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ποια ακριβώς θα είναι τα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τι βαθμό δηλαδή αυτά τα mega trucks, τα πιο μακριά και πιο βαριά φορτηγά, τι επιπτώσεις θα έχουν στο δικό δίκτυο της Ευρώπης. Η επιλογή λοιπόν για τα καταρχήν αποτελέσματα είναι το θέμα της ύπασης της ατμόσφαιρας, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όμως αυτό είναι ανεξάρτητο τελικά από την αιτία αυτή καθεαυτή της αλλαγής στον τρόπο μεταφοράς. Και εδώ υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μελέτες. Το θέμα του κόστους επίσης είναι πολύ σημαντικό. Αλλά στην ανάλυση κόστους οφέλους δεν την βρίσκουμε αρκετά στην μελέτη. Τόσο έχουν γραφτεί και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει το εξετάζουν το θέμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο φορές έχει εξεταστεί. Σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες που να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Άρα δύσκολα μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία. Γενικά μιλώντας λοιπόν, θα έλεγα ότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα της μελέτης είναι κάτι χρήσιμο αλλά από την άλλη μεριά χάνει κάπως το στόχο, το αντικείμενο για να φέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της από τη χρήση αυτή. Ένα άλλο ενδιαφέρον σενάριο που βλέπω εγώ είναι εκείνο των διαδρόμων όπου κάποιες χώρες μπορούν μεταξύ τους να συνονιθούν, να συζητήσουν και να επιτρέψουν μεταξύ τους ή σε κάποιους διαδρόμους μεταξύ τους να κυκλοφορούν αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, όπως έχουμε πει, με ταξιδίων χωρών καταρχήν. Είναι θεωρητική μελέτη αυτή βέβαια. Στην πράξη όμως οι πρακτικές εφαρμογές θα είναι μεγάλες και οι επιπτώσεις. Ευχαριστώ. In London. Keith, five minutes, please. Thank you and good afternoon. Ο Keith από το Λονδίνο. Θα κάνω μια γενική καταρχήν περιγραφή της αποτιμήσεις μου. Η μελέτη είναι χρήσιμη περιγραφή των προηγούμενων ερευνών που έχουν γίνει. Αλλά δεν είναι πλήρης. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Δεύτερον, δυστυχώς τα λεπτομερή συμπεράσματα και ιδιαίτερα τα σενάρια δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα προβλήματα που ταύτισε η ίδια η μελέτη. Τρίτον, αυτό που χρειάζεται για να μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις είναι μια πολύ λεπτομερέστερη έρευνα του, κατα... του λόγου για τον οποίο δεν υπάρχει συνένεση και τόσο πολλές διαφορές μεταξύ των μελετών. Τώρα οι λεπτομέρειες. Μερικά από τα θετικά στοιχεία τα ακούσατε και από άλλους. Πρώτον, δείχνει καλά τη σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ της cross elasticity και της εσωτερικής ελαστικότητας για τα φορτηγά συγκεκριμένα. Και είναι βασικό να καταλάβουμε την έννοια του αυτοκινήτου κάθετος χιλιόμετρων. Αυτά τα ξεχωρίζει καλά. Επίσης δείχνει καλά τις τρομερές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μελετών. Τώρα οι αδυναμίες της ταύτης Αμερικές και θα σας πω τις σημαντικότερες. Πρώτον, Πρέπει να συμπεριλάβουμε οπωσδήποτε και την επίπτωση της χρήσης των βαρέων φορτηγών, δηλαδή την μείωση της χρήσης των συνήθων φορτηγών. Ίσως αυτό να πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επόμενη οδηγία και αφορά και το περιβάλλον. Δεύτερον, οι αλλαγές του κόστους τόνου ανά χιλιόμετρο και όχι αυτοκινήτου ανά χιλιόμετρο. Τα αυτοκίνητα αυτά ταξιδεύουν μακρύτερα. Υπάρχουν και άλλες έννοιες βέβαια όπως τρόφιμα αναμίλη. Το θέμα είναι πώς το υπάρχον δίκτυο έχει όχι μόνο οικονομικές επιπτώσεις αλλά και περιβαλλοντολογικές στο κόστος. Άλλο θέμα που λείπει. Οι διαφορετικές αυτές μελέτες πρέπει να κάνουν τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικών μεταφορέων και εκείνων που είναι χοντρική μεταφορής. Η επιλογή ελαστικότητος είναι κάτι που έχει ήδη αναφερθεί. Η ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών μπορεί να είναι χαμηλή αλλά θα είναι ψηλότερη αν πάρουμε υπόψη μας το κριτήριο του τόνου χιλιόμετρο και του αυτοκινήτου ανά χιλιόμετρο. Η σουηδική μελέτη χρησιμοποιεί δεκαετή περίοδο στην οποία δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή στα συνήθη φορτηγά. Τη δεκαετία του 90 όπου συνέβησαν τέτοιες αλλαγές φάνηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν 20% λιγότερο οι σιδηρόδρομοι. Πρέπει λοιπόν και οι υπάρχουσες μελέτες να αναλυθούν λεπτομερέστερα. Τέλος, αφού δεν έχω χρόνο, για να καταλάβουμε γιατί δεν υπάρχει συνένεση και τόσο πολλές διαφορές πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα θέμα εσωτερικής εξοικονόμησης κόστους που δεν είναι το ίδιο με συνολική εξοικονόμηση κόστος, όταν λάβει κανείς υπόψη του δηλαδή και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κλπ. Η μείωση του εξωτερικού κόστους, δηλαδή το κόστος προς την κοινωνία ολόκληρη, είναι ο κύριος στόχος μας. Τέλος, δεν θα υπάρξει πρόοδος παρά μόνον όταν θα υπάρχει ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να μιλάει για αυτό το θέμα της κατανομής μεταξύ τρόπων μεταφοράς, τρένων και οχημάτων δηλαδή. Και αυτό να αποτελέσει μάλιστα μία δημόσια αποδεκτή λύση. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάω στους βουλευτές. Ε, έχουμε λοιπόν τους ε, βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Grosch, Mr. Alcadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr. Rike, Mr. Ertug, Mr. Benyon, Mr. Koch, Mr. Kramer. Okay. End of. No more putting... Μάλιστα. Τελείωσε λοιπόν. Κλείνω τον κατάλογο. Μην μου ζητήσετε το λόγο σε 45 λεπτά. Δύο λεπτά ο καθένα λοιπόν για να ακούσουμε και τι απαντήσει. Δύο λεπτά παρακαλώ και να ξέρετε ότι θα σα χρονομετρώ. Ξεκινάμε. Κύριε Γκρό, έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά, να ήθελα να σα ευχαριστήσω για την μελέτη, για την αξιολόγηση τη μελέτη και την εκτίμηση της μελέτης, ε, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συχνά ε, εξαρτάται και από τις προσδοκίες μας. Γιατί έχει και κανείς πολιτικές, ε, πολιτικές προθεσμίες, έχουμε την πίεση που ανεβαίνει, καταλαβαίνετε. Αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει σε πολλές περιστάσεις εδώ πέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι τότε είχαμε κάνει μια καλή πρόταση νομίζω να πούμε ότι καταρχάς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ένας γενικός κανόνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι η εφικτότητα αυτή, η οικονομική εφικτότητα που αναφέρατε, θα πρέπει να εξεταστεί από τον ίδιο το κλάδο. Ε, δεν φαντάζομαι αύριο μεθαύριο μια εταιρεία να πανεγοράσει ένα τέτοιο μεγάλο φορτηγό, αν δεν έχει κάτσει και έχει υπολογίσει ότι συμφέρει επόμενο σημείο στο οποίο συμφωνήσαμε. Δεν θα προωθήσουμε το δρόμο φρενάροντας παράλληλα θα προωθήσουμε τις οδικές μεταφορές φρενάροντας παράλληλα άλλους τρόπους ε, μεταφορών, αλλά δεν επενδύσουμε στους δρόμους, θα πρέπει να μην περιμένουμε και οικονομικά αποτέλεσμα. Έτσι έχει η κατάσταση. Άρα θεωρώ ότι αυτά που είχαμε συμφωνήσει τότε με την κυρία Γελασέντερ, να πούμε ότι το δημόσιος, ε, αν θέλει, το δημόσιος πληρώνει τις υποδομές, πληρώνει την ασφάλεια, πληρώνει όλα αυτά τα στοιχεία και αυτή η δημόσια διάσταση λοιπόν θα πρέπει να εκτιμήσει την κατάσταση από χώρα σε χώρα και να διαμορφώσει με ένα όμορφο τρόπο την κατάσταση. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελεί βάση για τη μελλοντική συζήτηση και ελπίζω να μπορέσεις, συνάδελφε, να συζητήσεις και μετά τις εκλογές την έκθεση αυτή επί της βάσης αυτής. Μάλιστα, ο κύριος Αλκαντράη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Βλέπω και τον συνάδελφο Λάιφριντ εδώ. Με τα ίδια δεδομένα καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα, ιδιαίτερα για αυτή την ελαστικότητα κατά πόσο θα μειωθεί ο αριθμός των ε, φορτηγών αντί να έχουμε μικρότερα λέμε να έχουμε μεγαλύτερα φορτηγά. Η ανταγωνιστικότητα όμως που αυξάνει στον τομέα των μεταφορών θα βάλει στη πάντα περισσότερα μέσα. Το ίδιο μπορώ να πω και για την ασφάλεια, ότι μεγαλύτερα φορτηγά, μεγαλύτερη όγκη και μεγαλύτερο βάρος θα έχει και μεγαλύτερες επιπτώσεις στις μεταφορές. Δεν ξέρω αν το έχουν κοιτάξει αρκετά οι μελέτες ποιες θα είναι ακριβώς οι επιπτώσεις και του κόστους με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να προσαρμοστούν οι μεταφορές στις νέες συνθήκες. Και στο τέλος, το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε περισσότερες οδικές μεταφορές ή θέλουμε να ενισχύσουμε μια πολιτική όπου έστω σε θελοντική βάση τα εμπορεύματα θα μεταφέρονται με άλλους τρόπους μεταφοράς και όχι ο δικός. Το υπογράμμισε και ο Γάλλος εμπειρογνώμων. Και έπειτα η Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 2005 δίνει κάποια φιλοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγούμε από τις οδικές μεταφορές. Τα εμπορεύματα δηλαδή να μεταφέρονται αλλιώς σιδηροδρομικά ή αλλιώς για μεγάλες αποστάσεις. Οπότε εγώ το θέτω ανάποδα. Σε τι βαθμό όλα αυτά που εξετάζουμε τώρα συνάδουν με τις φιλοδοξίες της Λευκής Βίβλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενιάν από τους φιλελεύθερους. Δεν έχουμε εδώ την κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ασφάλεια, βλέπουμε βελτίωση. Πώς όμως μετριέται με τους αριθμούς των ατυχημάτων ή των μοιραίων ατυχημάτων, γιατί ακούμε ότι μπορεί τα ατυχήματα να είναι πιο σοβαρά. Οπότε πώς υπολογίζονται αυτοί οι παράγοντες για να καταλήξουμε στην συνολική εικόνα. Εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα έπειτα. Με την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς τι γίνεται. Ε, 30 φορές λιγότερες είναι από ό,τι στις οδικές μεταφορές αν ακολουθήσουμε άλλα μέσα. Και τρίτον, τι γίνεται με τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης. Ο κύριος από τη Λουβέν το είπε. Είναι αλλιώς η εθνικές οδοί, αλλιώς η περιφερειακή, η αγροτική. Αν εγκριθούν τα μέγα τραξ για συγκεκριμένους διαδρόμους μεταφορών, όπως μας είπε, είναι κάτι άλλο. Από το να πούμε ότι απλώς απαγορεύονται από πολύ συγκεκριμένους δρόμους. Η μελέτη επίσης λέει ότι το κόστος αναβάθμισης των υποδομών κλπ. δεν μπορεί να το υπολογίσει. Αλλά και πάλι αυτό εξαρτάται από το μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε μια γενική έγκριση για τα φορτηγά αυτά, τότε φυσικά και θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις. Και έτσι έρχομαι και στο τελευταίο μου ερώτημα. Δεδομένου της δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη να συλλέξουν φόρους για ένα σωρό άλλα πράγματα που πρέπει. Αυτή η επενδυτική προσπάθεια πώς θα γίνει, σε τι χρονικό διάστημα περιμένετε να έχουν μαζευτεί τα χρήματα για τις επενδύσεις αυτές. Λίντεμπεργκερ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Την τελευταία φορά που το συζητήσαμε το θέμα αυτό και συζητήσαμε την μελέτη αυτή, μας προειδοποίησαν, νομίζω, μας προειδοποίησαν νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές που είχαν ασχοληθεί με το θέμα αυτό από την Επιτροπή μας ότι πέρα από την εφικτότητα, την οικονομική εφικτότητα θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ε, γενικότερη οικονομία των χωρών. Προφανώς τα πράγματα είναι διαφορετικά σε ορεινές περιοχές ε, ή σε, από τις άλλες περιοχές επίπεδες. Εξαρτάται και από το υπέδαφος. Το γεγονός όμως ότι δεν λάβαμε υπόψη τον παράγοντα αυτό, θεωρώ ότι είναι παράδεκτο. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα νέο μοντέλο κυκλοφορίας ε, μεταφορών. Να κοιτάξουμε δηλαδή τι σημαίνει όχι μόνο για την οικονομία των επιχειρήσεων, αλλά για την οικονομία των κρατών. Αναφέρατε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά είδατε τι θα γίνει με τα πάρκα, με τις πλατείες, με τις γέφυρες, τις σύραγγες που θα πρέπει να τραποποιηθούν. Τι κόστος συζητάμε. Κοιτάμε ορεινές περιοχές. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση αυτή. Είναι αδύνατον, αδύνατον. Άρα η μελέτη αυτή επιδεικνύει τεράστια χάσματα. Και να, επειδή αυτό το σημείο το οποίο είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή το κόστος που θα επιβαρύνει τα κράτη σε ό,τι αφορά το τρόπο μεταφοράς αυτής και σε ό,τι αφορά την επίδραση στους συνδρομικούς, ε, συνδρομικές μεταφορές μέσω της προώθησης ε, των οδικών μεταφορών, αυτά όλα λείπουν. Και με ενόχλησε το εξής. Μιλήσατε για τρεις ε, χώρες που έχουν εισαγάγει τέτοια φορτηγά και δεν έχουν καταργήσει ακόμα. Και εσείς από αυτό συμπεραίνετε ότι είναι ικανοποιημένες και ότι είναι καλά τα φορτηγά αυτά. Με τρεις χώρες ως βάση υπολογισμού θεωρώ ότι δεν είναι επιστημονικά αποδεκτά τα αποτελέσματα αυτά. Επίσης δεν υπάρχουν ε, επιστημονικά στοιχεία τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στις ε, μελέτες αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ρίκε. Δύο λεπτά. Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συντάκτες της μελέτης και να πω ότι τρία πράγματα ισχύουν για κάθε μελέτη που τα είπε και ο παρουσιαστής. Πρώτον, πολύ μεγάλη δυσκολία για να ληφθούν μέτρα για το σύνολο της Ευρώπης γιατί η δημογραφική, γεωγραφική, οικονομική σύνθεση της Ευρώπης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το Βέλγιο δεν είναι Σουηδία και η Ολλανδία δεν είναι Αυστρία. Δεύτερον, η οικονομική επίπτωση. Αν βάλουμε μεγαλύτερο όγκο και βάρος στα φορτηγά θα υπάρχουν μεγαλύτερες, περισσότερες εκπομπές και φυσικά περισσότερες οδικές σε σύγκριση με τις σιδηροδρομικές. Ένας ενδιαφέρον αριθμό είναι όπου και χρησιμοποιούνται τα βαρέα φορτηγά έχουν καταλάβει το 80% των οδικών μεταφορών. Τρίτον, η κοινωνικοπολιτική επίπτωση της χρήσης των βαρέων φορτηγών για τις ε, υποδομές είναι φανερή. Άρα θα χρειαστεί να αλλάξουν και ό,τι ισχύουν για τα πάρκινγκ κλπ. Τρίτον, για τα ατυχήματα. Τέσσερις φορές περισσότερα θύματα έχουν τα ελαφρά φορτηγά από ό,τι τα βαρέα. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω... Αυξάνονται μάλλον τα θύματα στα κανονικά φορτηγά, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μειωθούν από τα βαρέα. Συμπέρασμα, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικό, μόνο υποκειμενικό. Οι οικονομικοί παράγοντες στις μεταφορές είναι υπέρ των βαρέων φορτηγών, αλλά κοινωνικοπολιτικά το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα έπρεπε να το ξαναδούμε με μεγάλη φρόνηση. Χέρτσογκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω, μπορούμε να θεωρήσουμε μελέτη έναν κατάλογο copy-paste, αντιγραφής δηλαδή άλλων μελετών. Εμείς ως ε, Κοινοβούλιο πώς τη δώσαμε, πώς την αναθέσαμε αυτή τη μελέτη και με ποια κριτήρια επιλέξαμε τους εμπειρογνώμονες. Αυτό το ερώτημα να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ. Να περάσω και στα θέματα περιεχομένου. Ο κύριος Μακίδεν μίλησε για την έλλειψη στοιχείων, ότι είναι πολύ περιορισμένα τα αποδεκτικά στοιχεία. Γι' αυτό τα συζητάμε σήμερα αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε μελέτη αντικτύπου. Ύστερα ο Μακίνον είπε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, παροχές υπηρεσιών ε, στο σιδηρόδρομο. Έχουμε τη Λευκή Βίβλο, η οποία όμως τελικά δεν έχει εφαρμοστεί. Και αυτό να το συζητήσουμε. Να πω με πάσα ειλικρίνεια το εξή. Ε, στη μελέτη αυτή εξ αρχής θεωρούμε δεδομένο ότι θα μείνουμε στον τρόπο μεταφοράς των οδικών μεταφορών. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφορών όμως. Προφανώς λοιπόν θα υπάρχει αλλαγή τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών. Αν ξέρουμε ότι από σήμερα έως αύριο θα μειωνόταν 25 έως 30%, 30 το κόστος των οδικών μεταφορών, δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε καν ακόμα. Και κάτι που αυτό το αναφέρεται επιγραμματικά μόνο στη μελέτη σας. Να επανέλθω στο θέμα του κόστου. Στη Γερμανία και μόνο 11 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούμε μόνο για τις γέφυρες. Στην Αυστρία 5 ε, και πλέον ε, εκατομμυριά. Στην Πολωνία δεν αναφέρεται καθόλου τον Πολωνικό Υπουργείο. Και αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Και να πω επίσης, συνάδελφοι, ότι αυτή η μεταφορά στις οδικές μεταφορές θα σημαίνει ότι θα γίνουν ακόμα πιο φθηνέ οι οδικές μεταφορές και όλοι οι υπόλοιποι τρόποι πιο ακριβοί ή θα μείνουν εξίσου ακριβοί. Αλλά μια πρόταση, άλλη μια πρόταση, Πρόεδρε αυτά τα μεγάλα φορτηγά σε περίπτωση που τα επιτρέψουμε. Μου προκαλεί έκπληση που ναι. δεν ε, φωνάζουν και δεν διαμαρτύρονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις ε, θα ωφεληθούν γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σιγά που μπορούν να πληρώσουν και να αγοράσουν ένα τέτοιο φορτηγό. Πόσο μάλλον το λειτουργήσουν. Γι' αυτό λοιπόν να μας πει η Επιτροπή ποιος ε, έδωσε εντολή για την έκθεση αυτή. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Κοιτάξτε, να σας πω ότι δεν είναι τόσο κατανόητη η μελέτη αυτή. Πολύ απλά δεν ταιριάζει το συμπέρασμά τη σε κάποιο. Κοιτάξτε, γιατί μιλάμε για 60 τόνους, για φορτηγά 60 τόνων, για 40 τόνων. 44, 44 τόνων φορτηγά. Ας αφήσουμε τις σύραγγες, τους δρόμους, ε, τα τούνελ, τις γέφυρες, αν μιλάμε, εφόσον μιλάμε για 40 τόνους. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα, να μιλήσω για το μοντέλο. Δεν θέλω να έχω ένα πιο μεγάλο α, ε, όχημα απλό. Όχι, πιο μεγάλο, θέλω να δημιουργήσω ένα νέο σύστημα, ένα νέο μοντέλο με διαφορετικές ε, προδιαγραφέ, με διαφορετικό σύστημα πέδηση, με βιντεοκάμερες. Δεν θα... θα... Θα αντικατασταθούν έτσι τα παλιά φορτηγά και αυτό αναιρεί πάρα πολλά επιχειρήματα. Και τέλος, κοιτάξτε μία μελέτη στην Ερφούρτη που έγινε για την τεχνική ποικιλία για τη συνδυασμό μεταφορών μεταξύ φορτηγών και οδικών μεταφορών. Θα καταλήξετε σε διαφορετικά αποτελέσματα νομίζω στην περίπτωση αυτή κύριε Λάχιτβερτ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των φορτηγών αυτών, φυσικά πάντα σεβόμενοι την αρχή της επικουρικότητας. Ο κύριο Κράμερ, το μοναδικό θετικό για τη μελέτη είναι ότι αναφέρεται ότι οι διάφορες μελέτες δεν συμφωνούν ούτε για το φορτίο άξονα, ούτε για το κόστος, ούτε για τίποτα. Γιατί ο καθένας βρίσκει επιχειρήματα. Γι' αυτό και δεν μας βοηθάει όμως ε, η μελέτη αυτή. Και υπάρχουν μεγάλα κενά, για παράδειγμα, αυτά τα μεγάλα φορτηγά μιλάνε, ε, ενδείκνυνται για μεγάλες αποστάσεις που μπορεί να είναι συχνές αλλά όχι εδώ στην Ευρώπη. Να, να ζημιώσουμε δηλαδή, να ζημιώσουμε τις, τις δρομικές μεταφορές και να καταστρέψουμε τους δρόμους μας για να, να συγκρίνουμε τις υποδομές μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας που προσανατολίζονται σε τέτοιες υποδομές εδώ και χρόνια δεν χρειάζεται αλλαγή ουσιαστικά των υποδομών. Εμείς όμως χρειαζόμαστε τέτοια τροποποίηση γιατί για μας είναι κάτι καινούριο. Εδώ δεν έχουμε λεφτά στο Λεβερκούζεν και αλλού για να ε, φτιάξουμε και να επισκευάσουμε ήδη υφιστάμενες ε, γέφυρες. Δεν έχουμε χρήματα. Είναι τρελό αυτό που λέτε. Αναφέρθηκε το θέμα του κόστους. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δεν πρέπει να κινηθούμε. Αυτό που λείπει από την μελέτη είναι το Σε Μια μελέτη τον είπα ε, καταδεικνύει ότι 55% των συνδρομικών μεταφορών μεταφέρεται στους δρόμους. Αυτό είναι αντίθετο με κάθε αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ενώ ουσιαστικά δεν είναι συγκρίσιμο τίποτα. Δεν είναι συγκρίσιμο καν η... το δυναμικό που αξιοποιείται στα φορτηγά. Και φυσικά και κλείνω θα πρέπει να βελτιωθεί ε, η υποδομή όχι μόνο τα τούνη και οι γέφυρες αλλά κάθε ε, γωνία, κάθε στροφή και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Χέρτσοκ ε, τα κέρδη θα πάνε σε ιδιωτικά χέρια, ενώ ουσιαστικά η επένδυση θα έρθει από τα δημόσια κορβανά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Θα βάλω το χρονόμετρο. Και θα καταθέσω και τη δικιά μου άποψη. Εξετάζουμε την οικονομική πτυχή των μεταφορών. Αν μειώσουμε το κόστος των οδικών μεταφορών, ότι αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα οι σειροδρομικές μεταφορές να αναβαθμιστούν. Μα όποιος το λέει αυτό ζει νομίζω σε διαφορετικό κόσμο. Η προτεραιότητα της Επιτροπής μας είναι να αναπτύξουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδιαίτερα για τις εμπορικές μεταφορές να χρησιμοποιούνται οι σιδηρόδρομοι. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν το δρόμο των μεγάλων φορτηγών, mega όπως θέλετε τα λέτε, τότε αυτό που κάνετε είναι ότι στρεβλώνεται την αγορά και δυσκολεύεται ακόμα πιο πολύ του σιδηρόδρομου. Και κανένα δεν είναι πιο επικριτικό για του σιδηροδρόμους από μένα όσον αφορά τι αντιστάσει του ε, τι αλλαγέ κλπ. Γιατί πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία των ε, σιδηροδρόμων. Το δέχομαι αυτό, απόλυτα. Αλλά νομίζω ότι αν ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, τότε αυτό που κάνετε είναι ότι καταστρέφετε μια για πάντα τις εμπορικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου. Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος μου δεν είναι ότι αν επιτρέψουμε τα mega trucks ότι θα σταματήσουμε εδώ, μετά θα έχουμε τα ακόμα μεγαλύτερα. 60-72, εγώ νομίζω ότι έχουμε ακούσει όλα τα επιχειρήματα. Τότε τι θα πούμε πια. Γιατί θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το βάρος. Και γιατί υπάρχει αυτή η πίεση. Γιατί έτσι γίνονται πιο φτηνές οι οδικές εμπορικές μεταφορές. Αλλά αυτό δεν είναι το α και το ω της πολιτικής μεταφορών. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπε και η κυρία Λίχτεμπέργκερ, ότι υπάρχουν και κοινωνικές συνέπειες και δεν μπορείτε αυτές να τις αγνοήσετε επειδή οι οδικές εμπορικές μεταφορές γίνονται φθηνότερες. Λοιπόν, James, για να απαντήσετε και μετά στους αξιολογητές. Πέντε λεπτά εσείς και μετά λίγα λεπτά οι υπόλοιποι αν έχουν κάτι να προσθέσουν. Και δεν είσαστε υποχρεωμένοι να πείτε κάτι, αλλά η δημοκρατία επιβάλλει να σας δώσω το λόγο. James. Ε, πολλά ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά που μου απευθύνθηκαν προσωπικά. Ρωτήσατε πόσα μετριέται η ασφάλεια. Ε, αν είναι απλός αριθμός λιγότερων ατυχημάτων, όχι. Κάναμε την οικονομική αξιολόγηση της ασφάλειας, που σημαίνει το κόστος, τη σχέση μεταξύ λειτουργίας και ατυχήματος καθώς και του μεγέθους του ατυχήματος, όχι μόνο αριθμό θανάτων. Και ο λόγος που λέμε ότι μάλλον θα είναι θετική για την ασφάλεια η χρήση των βαρέων φορτηγών είναι ότι θα υπάρχουν λιγότερες κινήσεις οχημάτων. Πόσο συχνά θα είναι τα ατυχήματα και πόσο σοβαρά, ίσως σοβαρότερα αλλά λιγότερο συχνά. Επίσης ερωτήθηκε τι γίνεται όταν οι κυβερνήσεις δεν έχουν πολλά χρήματα για να αποζημιώσουν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι στη Σουηδία. Έβαλαν υψηλότερη φορολόγηση για τη χρήση των βαρέων στην Ολλανδία βασίστηκαν στην αντίληψη ότι κοινωνικά θα πλήρωνε το κράτος μόνο για την αύξηση του χώρου των σταθμεύσεων και όλα τα άλλα θα τα πλήρωναν οι χρήστες. Τι άλλο είχα... Ε, αν, δεν, αν βλέψαμε ορισμένα παράπλευρα κόστη. Όχι, όχι. Η μελέτη προσπαθεί ολόκληρο το κόστος να εξετάσει. Δεν παραγνωρίζει το δημόσιο κόστος για να κοιτάξει μόνο το ιδιωτικό κέρδος. Όλα τα κοιτάξαμε και την ασφάλεια και το περιβάλλον και αποσαφηνίζει ότι Υπάρχει μεγάλη διαφωνία και αβεβαιότητα. Δεν λέμε ότι υπάρχουν σαφείς και απλές απαντήσεις για όλα αυτά. Αλλά με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, που δεν είναι και πάρα πολλά, περιορίζονται στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση. Είπατε για τον πραγματικό κόσμο, μόνο στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν αυτά. Και εκεί φαίνεται ότι, από εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ωφέλη. Αλλά χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και αυτό το λέμε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να φανούμε ουδέτεροι. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε μονόπλευροι, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά των βαρέων, ούτε του ορέντη. Τα υπόλοιπα ίσως δεν ήταν ερωτήσεις αλλά σχόλια. Κοινωνικές πτυχές. για τις επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ποτίμηση, αλλά δεν είναι και ακριβής επιστήμη. Η ιδέα που είπε κάποιος ο, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί κατά του σιδηροδρόμου τότε θα έχουμε περισσότερες εκπομπές η έκθεση λέει ότι ο λόγος για τον οποίο θα υπάρξει μείωση μάλλον των εκπομπών είναι ότι υπάρχει λιγότερη εκπομπή ανατόνο από τα βαρέα. Εντάξει, δεν υπάρχει συνένεση και συμφωνία, το ξέρουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτά. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά τώρα για τους ε, reviewers μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε στην κλασική περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σχιζοφρένεια των μεν και των δε. Στη Γαλλία καταλήξαμε στο ότι αν αυξήσουμε την ταχύτητα στους δρόμους, ε, έχουμε επιπλέον θνησιμότητα. Παρόλα αυτά, ευτυχώς, η κυβέρνηση δεν αυξάνει την ε, ταχύτητα, γιατί το θέμα είναι συλλογικό. Οι εμπορικές μεταφορές, ακόμα και αν κάποιοι, κάποιοι θυμώσουν μαζί μου, τα εμπορεύματα μεταφέρονται δικός, καλός, εδώ και πολύ καιρό και θα παραμείνουν και οι εμπορικές μεταφορές ιδεοδρομικά θα παραμείνουν περιορισμένες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι περιορισμοί που μπαίνουν στις εμπορικές μεταφορές οδικός πρέπει να αυξηθούν. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί με το toll collect όπως γίνεται στην Γερμανία, ελπίζω να γίνει και στη Γαλλία. Για να κερδίσουμε σε ασφάλεια αυτό που λέμε για την ασφάλεια με τα mega trucks ότι θα μπορούν οι οδηγοί να καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τι συμβαίνει και στο μπροστινό μέρος και στο πίσω μέρος του φορτηγού, στο αξόνι κλπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι περισσότερη ασφάλεια. Και όχι να προσπαθούμε σών και καλά να επιβάλλουμε τα Megatrax. Πρέπει να προσπαθούμε να επιβάλλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια των φορτηγών στους δρόμους μας Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί έχω εμπειρία από τη χιλία της Ηνωμένες όπου κάθε τόσο σταματούν για να ελεγχθεί το βάρος του φορτίου τους τα φορτηγά στους δρόμους. Κάθε τρεις και λίγο χωρίς διαμαρτυρίες. Ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Μακίναν. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με όλες αυτές τις εταιρείες, πολλές στην Ευρώπη, που δεν έχουν την επιλογή να επιλέξουν. Εξαιτία των προϊόντων που μεταφέρουν ε, και άλλων ε, παραγόντων πρέπει οδικά να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν αυτές οι εταιρείε και θέλουν είναι βελτίωση των οδικών τους μεταφορών. Δεν πρόκειται να καλυφθούν πολλές εμπορικές μεταφορές, χαμηλής πυκνότητας για παράδειγμα. Αυτό το οποίο περιορίζει την κατάσταση είναι πιο πολύ ο τρόπος με τον οποίο ε, φορτώνονται τα φορτηγά αυτά που είναι κυβικού τύπου. Οι μελέτες, μελέτες που αξιολογήθηκαν είναι μελέτες με σενάρια που εξετάσουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Τη σημερινή συζήτηση επικεντρωθήκαμε στα 25 μέτρα 60 τόνοι. Αλλά δεν θα έπρεπε. Αν έχουμε φορτηγά τα οποία έχουν το ίδιο βάρος με αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά που η κυβική τους χωρητικότητα αυξάνει, αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Γιατί όντω άμα είναι πιο βαριά χρειάζονται καινούριε γέφυρε, καινούρια τούνελ, ενώ στην άλλη περίπτωση όχι. Και μετά πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πρόσβαση των φορτηγών αυτών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τηλεματική, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την μετακίνησή τους ή μπορούμε να πούμε σε ποιους δρόμους θα επιτρέπονται αυτά τα φορτηγά, ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις επί των υποδομών. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά δηλαδή, γιατί εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε από τα διέξοδο. Όσο βέβαια εξετάζουμε ένα είδο μόνο φορτηγών και πάντα τα συγκρίνουμε με του σιδηρόδρομου, δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Ευχαριστώ, κύριο Μπρίμε. Έχω μια γενική παρατήρηση είναι πολύ μικρή η πιθανότητα σύντομα να μειωθεί η οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Και όλοι προσπαθούν την παραγωγικότητά τους να την αυξήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Τα μεγάλα αυτά φορτηγά είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η παραγωγικότητα σε αυτό το τομέα αλλά και οι σιδηρόδρομοι και άλλες ε, μορφές μεταφορών προσπαθούν να πετύχουν αύξηση. Αυτή είναι μια σκέψη που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο κύριος Βακάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σημεία. Πρώτον, κι εγώ είμαι οικονομολόγος ειδικευμένος στις μεταφορές είναι γνωστό ότι οι οδικές μεταφορές έχουν μεγάλο εξωτερικό κόστος. Αν λοιπόν μειωθεί το εσωτερικό κόστος, τότε το κοινωνικό κόστος είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί. Αναφέρθηκε και νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουμε απόψη μας στην όποια απόφαση. Δεύτερον, το θέμα του βάρους και του μεγέθους. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία όσον αφορά την κυβική διάσταση και το βάρος. Αν σχεδιαστεί ένα τέλειο φορτηγό όσον αφορά τον όγκο του, εξορισμού, δεν θα είναι καλό για κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν περιορισμούς όσον αφορά το βάρος και θα πούν ότι όχι, πρέπει να αλλάξει για να ταιριάζει καλύτερα στις δικές μας τις ανάγκες. Θα υπάρχει δηλαδή μια συνεχής πίεση. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε σαν επαγγελματίες του κλάδου. Τέλος, κάτι που δεν αναφέρθηκε αρκετά, αλλά είναι πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη και αυτό είναι η τιμή για να λύσουμε το ζήτημα. Αν λοιπόν πούμε ότι θα μειώσουμε το εσωτερικό κόστος, των ε, φορέων και χρησιμοποιούμε περισσότερο μεγάλα φορτηγά. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε όλες τις μελέτες. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν κατανοητά και να καταλάβουμε ότι χρειάζεται ο συνδυασμός του εξωτερικού και του εσωτερικού κόστους για να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η συζήτηση και θα μιλήσω αγγλικά γιατί δεν είναι πλέον τόσο τεχνικά τα ζητήματα, τόσο περίπλοκα. Να ζητήσω συγγνώμη που ήμουν τόσο αυστηρό ε, στην αρχή, αλλά από πλευρά περιεχομένου νομίζω ότι θα μείνω στην αρχική μου εντύπωση. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι ήταν τόσο διαφορετικές και διστάμενες οι απόψεις των ε, εμπειρογνωμόνων. Δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα σε σχέση με πριν. Είπαμε στη μελέτη ότι όλα είναι πιθανά και δυνατά. Δεν έχουμε κάποιο έγγραφο στο οποίο να μπορούμε να βασίσουμε την απόφασή μας και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στην Επιτροπή Πώς θα συνεχίσουμε από τώρα. Θα ήθελα μία μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το ήθελα αυτό. Το ομολογώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβιάστηκε. Δεν είχαμε τη μελέτη αντικτύπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη και ιδιαίτερα στη συζήτηση που ακολούθησε. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τι λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Στυρ, τη Στυρ Ντέβις και τους τέσσερις εμπειρογνώμονες που αξιολόγησαν τη μελέτη, Κρόιζε, Μακίνεν, Πρίσοβεσον και Μπάκιν για τις παρεμβάσεις τους. Ξέρω ότι ήταν πολύ συνοπτική συζήτηση, ήταν όμως απαραίτητη να σας πω το εξής φεύγοντας ε, και προς τους εμπειρογνώμονες. Δεν έχω πιστεί γιατί χρειαζόμαστε μεγάλα φορτηγά όταν τα φορτηγά που χρησιμοποιούμε είναι τέλεια στις μεταφορές. Και μάλιστα πολλές φορές ε, κυκλοφορούν και άδεια. Νομίζω ότι πιο πρακτικό θα ήταν και πιο αποτελεσματικό να φροντίσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα φορτηγά που έχουμε στη διάθεσή μας και να μην κυκλοφορούν άδεια. Σας ευχαριστώ όμως για τις απόψεις σας. Όπως βλέπετε το θέμα αυτό προκαλεί έντονα συναισθήματα και έντονες αντιδράσεις ε, στους βουλευτές. Όλοι νοιάζονται ιδιαίτερως για το θέμα αυτό, είναι να το πω και ήπια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, δύο λεπτά διάλειμμα και μετά προχωράμε στο επόμενο θέμα.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 Okay, can we get started? Ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Παρακαλώ τους εμπειρογνώμονες να έρθουν να καθίσουν εδώ, δίπλα μου. Παρακαλώ, όσοι δεν θα παραμείνετε εδώ για το θέμα του τουρισμού, τη συζήτηση τρογγυλής τραπέζι δηλαδή που θα κάνουμε, τότε παρακαλώ αποχωρήστε. Όσοι πάλι είναι για αυτό το θέμα, παρακαλώ καθίστε και οι πυρογνώμονες να έρθουν εδώ δίπλα μου. So the next point on the agenda... Επόμενο θέμα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση στον Αγγλής Τραπέζης με θέμα τουρισμός για όλους. Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός σήμερα στην Ευρώπη σχετικά με την εποχική του διάσταση και την πρόσβαση στον τουρισμό. Έχουμε εδώ τον ε, προεδρεύοντα για την ε, συζήτηση αυτή που θα κάνουμε από την Αγίδα της Επιτροπής μας. Έχουμε και πέντε εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέμα της εποχιακότητας και της πρόσβασης στον τουρισμό. Έχουμε τον κύριο Ρομπέρτο Βιτάλη που είναι πρόεδρος της Ιταλικής Οργάνωσης Village for All. Έχουμε την Αν Χέρμανς που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας AIDS τον Άννη Σίλβα που είναι συντονιστής του προγράμματος Εκαλύψω για το Ίστο που είναι κοινωνικός ε, τουρισμός, ο Πάλο Μπονίνη που είναι πρόεδρος του Νέστουρ και τον Εδουάρδο Σανταντέρ που είναι ε, διευθυντής της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Ταξιδιού. Η κυρία Τουντίνη είναι επίσης εδώ και η κυρία Καρέρα από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Καλό. Πέντε λεφτά εισαγωγή και μετά πέντε λεφτά εμπειρογνώμονες και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Κάρλο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε όλοι. Αρχίσαμε τις εργασίες της Task Force για τον τουρισμό μέσα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού με προπαρασκευαστικά έγγραφα. Και προσπαθήσαμε να έχουμε την κατάλληλη στιγμή και αυτή τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για να δούμε πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, η οποία αναφέρεται και ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε με την έκθεση πρωτοβουλίας μας που εγκρίναμε τον Οκτώβριο του 2011. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του σενάριου καθορίσαμε τις προτεραιότητές μας και σήμερα συζητάμε για την πρώτη από αυτές τις προτεραιότητες και επιλέξαμε δύο θέματα που έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Είναι το θέμα της εποχιακότητας και το θέμα της πρόσβασης, της προσβασιμότητας, πώς δηλαδή θα έχουν όλοι πρόσβαση στον τουρισμό είναι και κάτι επίγον για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Έχουμε διαπιστώσει πως όλοι οι φορείς του τομέα διαπιστώνουν πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους πέρα από τους δύο μήνες που είναι η κλασική περίοδος η τουριστική. Άρα λοιπόν το θέμα της εποχικότητας έχει μεγάλη σημασία. Πώς δηλαδή θα επιμικίνουμε την τουριστική περίοδο. Είναι μια μεγάλη προτεραιότητα αυτή, έτσι το θέτουν όλοι οι τουριστικοί φορείς. Έπειτα, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν 80 εκατομμύρια περίπου Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν κάποια αναπηρία και άρα έχουν ειδικέ ανάγκες για να έχουν πρόσβαση στον τουρισμό, όπως και οι οικογένειες με μικρά παιδιά, έτσι. Αλλά υπάρχουν και όλες αυτές οι περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό λοιπόν και σκεφτήκαμε ότι χρειάζεται μια ειδική πλατφόρμα που να βοηθήσει τις περιπτώσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο, είναι ηθικό για να μπορούν να είναι τουρίστες, να αποφελούνται από τον τουρισμό όλοι. Από την άλλη μεριά σκεφτόμαστε ότι είναι και χρήσιμο οικονομικά μιλώντας για τις επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο λοιπόν στοιχεία μαζί μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην προσβασιμότητα στον τουρισμό για όλους και ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για να περιορίσουμε τις διακρίσεις και να ενισχύσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και θέλουμε λοιπόν και αποφασίσαμε να προωθήσουμε αυτή τη συνάντηση που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας και να μπορέσουμε να ακούσουμε τις διάφορες απόψεις από όλους τους φορείς που είναι σήμερα εδώ παρόντες. Έτσι θα δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση αυτή που έχει ξεκινήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κλείνω λέγοντας ότι δεν ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό της πρόσβασης στο τουρισμό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί για τρίτο χρόνο ουσιαστικά, κάτι το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει εδώ και ο πρόεδρος. Γι' αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόρους και ξέρουμε ότι ήδη χρησιμοποιεί για να ενισχύσει την πολιτική αυτή. Άρα λοιπόν ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει πριν από τρία χρόνια και θέλουμε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες λοιπόν και μετά θα ακούσουμε και τους ε, συναδέρφους που σίγουρα όλοι έχουν να αναφέρουν σημαντικά θέματα. Thank you very much. If I start off then with Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ρομπέρτο Βιτάλη, πρόεδρος της οργάνωσης Χωριό για Village for All. Παρακαλώ κύριε Βιτάλη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής που οργανώσατε τη σημερινή συνάντηση. Η οργάνωση Village for All είναι μια οργάνωση που θέλει να δημιουργήσει φιλοξενία για όλους. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού, την ΕΝΙΤ, και της εταιρείας ε, στην οποία ανήκουν ε, τα κάμπινγκ. Υπό την αιγίδα λοιπόν αυτών φτιάξαμε την οργάνωσή μας. Ανήκουμε στην WO και της οργάνωσης των managers στον χώρο του τουρισμού και είμαστε και μέλη της ΕΝΑΤ που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόσβασης στον Τουρισμό όπου συμμετέχουν οι επαγγελματίες του τουρισμού. Γι' αυτό και χαιρετίζω εδώ και την Άννα Γκράσια Λάρο που είναι πρόεδρος και που θα ήθελε να είναι εδώ σήμερα, αλλά δεν μπορούσε για να συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Αποστολή μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε την ευκαιρία για διακοπές για όλους. Να μπορούν όλοι να συμμετέχουν είτε πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά, είτε πρόκειται για άτομα με αναπηρίες, είτε πρόκειται για ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ασθένεια, για τους ηλικιωμένους. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα άτομα στον, για όλα αυτά τα άτομα στον τουρισμό. Και αυτό το κάνουμε μέσω ενημέρωσης πρώτα απ' όλα, για να ενημερώσουμε τους πελάτες αυτούς να βελτιώσουμε το επίπεδο προσβασιμότητας των ατόμων αυτών, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές για την ε, προσβασιμότητα στον τουρισμό. Εξάλλου ο καθένας έχει ειδικέ ανάγκες. Θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση λοιπόν και να δημιουργήσουμε αυτό το πνεύμα της φιλοξενίας που να τα αποκρίνεται στις ανάγκες όλων και στις ειδικέ ανάγκες των ειδικών αυτών πελατών όταν θέλουν να πάνε διακοπές. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε έναν κατάλογο με τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να βελτιωθούν. Αυτό είναι ο στόχος μας. Γιατί οι δομές που πιστοποιούνται από εμά ελέγχονται κάθε χρόνο και συνεχώς ζητάμε να βελτιώνουν την προβασιμότητά τους. Λειτουργούμε στην Ιταλία και στην Κροατία και πολύ σύντομα και στη Βραζιλία, στις χώρες Μπενελούξ, στο Ενωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Το σύστημα με το οποίο δουλεύουμε είναι τέτοιο που δημιουργήσαμε την, ε, το app V4A που προσπαθεί να απαντήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων και να μην ακολουθήσουμε μια τυπολογία, κάποιες προδιαγραφές δηλαδή γενικές. Το σύστημά μας, η μέθοδός μας, δημιουργεί ένα σύστημα πληροφορικής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τις εθνικές προδιαγραφές. Θέλουμε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συγκεκριμένων καταναλωτών και τους ενημερώνουμε για να μπορούμε και να τους βοηθήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε τα όσα αναφέρει και ο κώδικας ε, δεοντολογίας που έχουμε στο Βένετο, αλλά και άλλες συμβάσεις για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για παράδειγμα. Και έτσι προσπαθούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά το κύριο σημείο αναφοράς μας είναι βέβαια η Ευρώπη προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιτάλη. Τώρα η κυρία Αν Χέρμανς για την Age Platform Europe. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, αξιότιμη βοηθή και προσκεκλημένη. Χαίρομαι που συμμετέχω εδώ σήμερα και θα σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις από την εμπειρία μου. Καταρχάς, η, η πλατφόρμα της Ευρώπης, ε, μια ε, οργάνωση ομπρέλα που περιλαμβάνει αυτή η οργάνωση AGE Platform Europe, διάφορες άλλες οργανώσεις. Ε, θα σας αναφέρω λοιπόν στο κείμενο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τουρισμό για τους ε, ηλικιωμένους... και ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, προετοίμασα μια παρουσίαση, την οποία και θα συνοψίσω όμως τώρα σε κάποια σημεία κλειδιά. Καταρχάς, διαπιστώνουμε σε ευρύ επίπεδο παγκοσμίω ότι οι ηλικιωμένοι αυξάνονται και οι πιο πολλές οργανώσεις οι τουριστικές προσανατολίζονται στους νέους ηλικιωμένους, αν θέλετε, στους ηλικιωμένους που είναι ακόμα υγιείς. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Και είναι, αν θέλετε, και πιο η κλασική ομάδα στην οποία α, απευθύνονται οι τουριστικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις, λαμβάνοντας υπόψη και ότι, για παράδειγμα, αυτή η ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο, προτιμά τα ταξίδια και, για παράδειγμα, έχει κάποιες προτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με πλοίο. Επίσης, σε ό,τι αφορά και τον τουρισμό στην περιοχή του καθενός. Ο τουρισμός είναι Αφενός ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται από τη ζήτηση ανάλογα με την αγορά, αλλά φυσικά παίζουν ρόλο και τα διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης, διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προωθήσουν συγκεκριμένα είδη τουρισμού σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον τουρισμό που είναι φιλικός προς τους ηλικιωμένους. Στην ε, ομάδα αυτή των ηλικιωμένων που έχουν δικαίωμα στον τουρισμό υπάρχουν και μια ομάδα που έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά θέματα υγείας, θέματα ευεξίας, κάποιες διακοπές ε, για συγκεκριμένη φροντίδα, αλλά και ο τουρισμός για όλους. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, αν θέλετε, στην γενικότερη προσβασιμότητα, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στον τουρισμό και όλοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τουρισμό. Αλλά παράλληλα αυτά υπάρχουν κάποιες ε, συγκεκριμένες οργανώσεις που χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι θα πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση και να φροντίσει πραγματικά όλοι να έχουν πρόσβαση στον τουρισμό και να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές στο βαθμό του δυνατών του δυνατού και βλέπουμε ότι κάποιες οργανώσεις έχουν για παράδειγμα ηλικιακό όριο για τις ε, ασφάλειες. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει την προσβασιμότητα αλλά και την βιωσιμότητα. Γιατί οι ηλικιωμένοι δεν είναι αυτονόητο, αλλά χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται στα σημερινά ερωτήματα. Ε, θα πρέπει να συμμετέχουν και πιο πολύ στην πολιτική, στη χάραξη της πολιτικής. Αυτό αναφέρεται σε διάφορα κείμενα. Χαίρομαι, χαίρομαι που αναφέρεται και θα ήθελα πραγματικά αυτό να γίνει στο μέλλον. Οι ηλικιωμένοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν, να σε αυτές τις ε, πολιτικές. Ελπίζω επίσης η πολιτική να συντονιστεί λίγο, προκειμένου να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των πιο ηλικιωμένων. Και έτσι η Ευρώπη να μην είναι μόνο πρώτη στην παροχή τουριστικών τέτοιων υπηρεσιών, αλλά και στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών φιλικών προς τους ηλικιωμένους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάνι Σίλβερ, συντονιστής project ε, της Διεθνούς Οργάνωσης για τον Τουρισμό. Έχετε πέντε λεπτά της ε, οργάνωσης e Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την που έχει δημιουργήσει την έννοια, την ιδέα της προσβασιμότητας όλων σε διακοπές στον τουρισμό. Η βασική μας έννοια τα 50 χρόνια που υπάρχουμε είναι όχι μόνο να δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στον τουρισμό αλλά και να στηρίξουμε τον τουριστικό τομέα με την προσβασιμότητα σε όλους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες του Ίστο είναι να γνωστοποιήσουμε την έννοια του κοινωνικού τουρισμού, να προωθήσουμε πιέσεις για ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και υποστήριξη της διευκόλυνσης των διακοπών για όλους. Τα πρόσφατα χρόνια τους τελευταίους μάλιστα μήνες θα έλεγα, αναλήφθηκε μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Κομισιόν, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, το σχέδιο Καλυψό. Ή μάλλον το σχέδιο Εκαλύψ. σε συνδυασμό με την πολιτική αλλά και την πρακτική πλευρά της οργάνωσής μας, ταυτίσαμε το γεγονός ότι ο τουρισμός εξαρτάται εμπολής από τον ιδιωτικό τομέα και το έκαλυψ θέλει, στοχεύει ιδιαίτερα στους πιο ηλικιωμένου, στους αναπήρους, τους νέους και γενικά τους ανθρώπους με δυσκολίες. Οι συγκεκριμένες αυτές αγορές μέσω του προγράμματος Εκαλύψ έχουν έναν τρόπο, μια πρόσβαση για τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων τουρισμού αλλά και περισσότερη πληροφόρηση. Αυτό αφορά βέβαια και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τις δραστηριότητε μας για αυτές τις ηλικιακέ και άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Αυτό το θέμα του συνδυασμού δύο τομέων μας προέκυψε από την ανάγκη να υπάρξει μία πιο πανευρωπαϊκή έννοια κοινωνικού τουρισμού. Συνήθως τον κοινωνικό τουρισμό τον βλέπαμε ως μεμονωμένη εθνική πρωτοβουλία ενώ τώρα θέλουμε να γίνει ενωσιακή μέσω του ΕΚΑΛΥΠΣ διότι ανακαλύψαμε ότι κάθε χώρα της Ένωσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναλαμβάνει δραστηριότητες μεμονωμένα που βασικά συμφωνούν με τις αρχές μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το εκαλύψ ώστε να δώσουμε τις ίδιες δυνατότητες σε όλους, δηλαδή ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ένα θέμα διακοπών και διασκέδασης αλλά και μάθησης και παιδείας. Μέσω του εκαλύψου λοιπόν και με βάση μη κερδοσκοπική θέλουμε να βελτιωθεί και η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα αλλά και η πρόσβαση σε εκείνες τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν. Potential points that we must άλλα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Ίστο. Εμείς θεωρούμε, επειδή είμαστε διεθνής οργάνωση, ότι υπάρχει ε, πανευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή, γενικά, οι δραστηριότητες του κοινωνικού τουρισμού παρέμεναν εθνικές μέχρι πρόσφατα. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές χώρες μέλη, ότι υπάρχουν οργανώσεις, ιδρύματα που χορηγούν υπηρεσίες κοινωνικού τουρισμού αλλά πάντοτε παραμένουν σε χώριο επίπεδο ενώ σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη θέληση και ενδιαφέρον όχι από, από την Ίστο αλλά και από άλλους παράγοντες του κοινωνικού τουρισμού μια θέληση να ξεπεράσουν τα εθνικά σύνορα, να ανακαλύψουν οι κοινωνικοί τουρίστες και νέες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τώρα ο κύριος Πάολο Μποντζίνη, πρόεδρος του Next Tour Βρυξελών. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνεται στην οργάνωσή μας να έρθει εδώ. Πρέπει να πω ότι το δικό μας το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει, χρηματοδοτείται. Είναι ένα δίκτυο τουριστικών περιοχών και μιλάμε εδώ για την περιοχή της Τοσκάνης. Αλλά συμμετέχουν και η Καταλωνία και άλλες περιφέρειες. Εκεί που υπάρχει πολλής τουρισμός. Συνολικά είμαστε 27-28 περιφέρειες. Υπάρχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και πανεπιστημιακοί. 30 πανεπιστήμια συμμετέχουν στο δίκτυό μας. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο δίκτυο, σε θελοντική βάση είναι η συμμετοχή και ετησίως όσοι συμμετέχουν πληρώνουν κάτι. Είναι ένα δίκτυο λοιπόν το οποίο δίνει μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητα. Με την ευρή έννοια του όρου. Πρώτα απ' όλα φροντίζουμε να προσφέρουμε στην επόμενη γενιά ένα κόσμο που θα έχει προστατεύσει τους σπόρους, τις πηγές και σε αυτά τα πλαίσια να βλέπουμε τον τουρισμό. Πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι η θεματική μας, τα θέματά μας δηλαδή, τα βλέπουμε ως εξής. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο τουρισμός είναι ένας τουρισμός που να ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη τυπολογία και θα χρησιμοποιείται για να ξεφύγουμε από το έλλειμμα μια συγκεκριμένη σεζόν. Όχι, δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο δίκτυό μας, το Nexto, είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τα πιο σημαντικά στοιχεία που για μας είναι ο κοινωνικός διάλογος πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, επί τόπου πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις του πληθυσμού. Δηλαδή, ο ίδιος ο πληθυσμός τι είδους τουρισμό θέλει στην περιφερειά του. Θέλουμε δηλαδή να υπολογίσουμε πολλά και διάφορα πράγματα. Υπάρχει το θέμα του περιβάλλοντος, υπάρχει το θέμα των αποβλήτων, υπάρχει το θέμα της ενέργειας, αλλά υπάρχει και το θέμα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής που δεν πρέπει να υπονομεύεται από την παρουσία τουριστών. Μπορούμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες αν θέλετε, αλλά εμείς έχουμε αναπτύξει διάφορους δείκτες. Γιατί το Next Tour, το δίκτυό μας, στην ανακοίνωση της Επιτροπής 352 του Ιουνίου νομίζω το 2010, στη δράση 11, το Next Tour είναι το δίκτυο το οποίο καλείται να αναπτύξει μοντέλα διαχείρισης προορισμών υπέρ του βιώσιμου τουρισμού. Η διαφοροποίηση πρώτα απ' όλα μέσα σε όλη τη χρονιά και να μην ε, συμπιέζεται ο τουρισμός μόνο ένα-δύο μήνες το χρόνο, αλλά αυτό να γίνεται σεβόμενη την ποιότητα της ζωής του πληθυσμού επιτόπου. Mm. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους ανα πάσα στιγμή. Να μην είναι εποχιακός. Υπάρχουν ε, περιφέρειες που έχουν προγράμματα ακριβώς για να μην είναι ο τουρισμός εκεί εποχιακός. Υπάρχουν περιοχές που ασχολούνται περισσότερο με το θέμα της προσβασιμότητας. Οπότε επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μερικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που έχουμε. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν πως κάποιες περιοχές μέσω των προγραμμάτων τους αυτών που υποφελούνται από κοινοτικά κονδύλια έχουν προχωρήσει. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να μπούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Εντουάρτο Σανταντέρ που είναι διευθυντής της CTC. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και για όσοι δεν μας γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Ταξιδιών είναι μια ε, οργάνωση ομπρέλα που έχει το σκοπό να ε, προωθήσει τις υπερατλαντικές, τα υπερατλαντικά ταξίδια. Η Ευρώπη παραμένει ο πρώτος ε, προορισμός για τους τουρίστες το 2012 πρέπει να σας πω ότι είχαμε 52% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Παρά το γενικά αρνητικό οικονομικό κλίμα σε συνδυασμό με το συνδρομή του κλάδου στο ΑΕΠ των χωρών καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι ο τομέας του τουρισμού και υπογραμμίζει την σημασία του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανταγωνιστικότητα έχει να κάνει με την βιωσιμότητα του τουρισμού, προκειμένου να υπάρχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και δεοντολογικά ζητήματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις περιφέρειες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικο-πολιτισμικά ζητήματα καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Γιατί λοιπόν η Επιτροπή μας προασπίζει τον βιώσιμο τουρισμό. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά αλλάζουν αν θέλετε και οι τρόποι τουρισμού. Υπάρχει για παράδειγμα ο τουρισμός για όλους. Ένα δισεκατομμύριο ε, άνθρωποι στον κόσμο υπολογίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ζουν με κάποια αναπηρία. Μαζί με τα με, μέλη της οικογένειάς τους, λοιπόν, μιλάμε για το 1 τρίτο, μάλλον συγγνώμη, για 15% ε, του πληθυσμού. Ένα στους τέσσερους, τέσσερις Ευρωπαίους υπολογίζεται. Έχει κάποιον στην οικογένειά του με κάποια αναπηρία. Επίσης υπάρχουν κοινωνιοδημογραφικές αλλαγές στην σύσταση του πληθυσμού και αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο ταξιδίων και αυτό θα επηρεάσει τις αγορές αυτές. Θα επηρεαστούν, για παράδειγμα, η Κίνα αλλά και η ΙΠΑ και ο Καναδάς που είναι καθιερωμένες αγορές. Επίσης, η εποχικότητα επηρεάζει το 96% και πλέον των προορισμών. Αυτό φυσικά επιβαρύνει όλες τις δομές, επίσης η ελαστικότητα των τιμών στα τουριστικά μέρη. Προωθούν την διαφοροποίηση και την ποικιλία των ε, παροχών προκειμένου να περιλαμβάνουν για παράδειγμα φεστιβάλ, εκδηλώσεις και το καθεξής. Άρα η προσβασιμότητα και η εποχικότητα είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και η μεσαία η οποία αυξάνεται στον αριθμό της ζητά λοιπόν τέτοια πρόσβαση και μάλιστα με τρόπο περιβαλλοντικά και πολιτισμικά φιλικό θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Αυτά λοιπόν είναι φιλοδοξίες. Πέρσι λάβαμε ένα εκατομμύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους αυτούς. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ορόσημο για την ETC. Γιατί θα πρέπει να καθιερωθεί ακόμα πιο πολύ η Ευρώπη στο παγκόσμιο προσκήνιο. Χρειαζόμαστε τρία στοιχεία. Καταρχάς, είναι βασικό οι εθνικές οργανώσεις τουρισμού να ενισχύσουν την συνεργασία τους, αναπτύσσοντας μια ευρωπαϊκή ταμπέλα, αν θέλετε, κατά δεύτερον, να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και τρίτον, βαθιά συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε η κυρία Φραντσέσκα Τουντίνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στο εργαστήριο αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Με παρακάλεσαν να σας αναφέρω ποιες δραστηριότητες έχουμε στα πλαίσια της ε, βιωσιμότητας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσω να σας παρουσιάσω το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Θα είμαι σύντομη λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι βιωσιμότητα και η στοχοθεσία των δραστηριοτήτων. Εμείς σίγουρα έχουμε στο στόχαστρο, έχουμε στο επίκεντρο των προσπάθειών μας ε, την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η προσβασιμότητα. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας ε, έδωσε και η πρωτοβουλία Εκαλύψ μας έδωσε νέες Καλύψω. μας έδωσε νέες ε, προσδοκίες, νέες ε, δυνατότητες σε ό,τι αφορά τις τουριστικές ροές μεταξύ των κρατών μελών που θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε ενδεχομένω. Μέχρι τα τέλη του έτους θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε έως και τέσσερα projects σε 30.000 ε, με 30.000 ευρώ το κάθε project και θα δούμε τι θα καταφέρουμε. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά προϊόντα, σε ό,τι αφορά την βιώσιμη κατανάλωση και επίσης για τις ε, εποχές ε, που δεν έχουν υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες. Ο Επιτροπός Ταγιάννη έκανε διάφορες πολιτικές συμφωνίες με διάφορες χώρες. Τις πιο σημαντικές χώρες, για παράδειγμα, BRICS, για να προωθήσει και να ενισχύσει τις τουριστικές ροές. Και εισάγαμε ένα πρόγραμμα πιλωτικό με 50.000 τουρίστες με τη Λατινική Αμερική για να προωθήσουμε τον τουρισμό σε μη ε, σε μη high season, αν θέλετε, σε εποχές που δεν έχουν πάρα πολλούς ε, νεκρές ε, περίοδους. Στο στόχο λοιπόν, βάζουμε το θέμα της προσβασιμότητας και Έχουμε φυσικά και στο επίκεντρο τον τουρισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ασχολούμαστε με θέμα της χορήγησης, ε, για παράδειγμα, θεωρήσεων. Ασχολούμαστε με τους ταξιδιώτες ε, που χρησιμοποιούν αεροδρόμια. Δεν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στους τουρίστες με αναπηρία. Τα θέματα λοιπόν αυτά έχουν να κάνουν με την αρχή ότι η Ευρώπη πάντα είναι ανοιχτή και διτεθειμένη να καλωσορίσει τους επισκέπτες και έχουμε κάνει και μια διαφήμιση σε παγκόσμιο επίπεδο όπου αναφέρουμε ότι η Ευρώπη έχει τέσσερις εποχές και πάντα σας καλωσορίζει. Σε αυτά λοιπόν θα περιοριστώ και αν θα απαντήσω και ερωτήσεις άμα χρειαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρος. Η Καρέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω το πανόραμα. Πώς χρησιμοποίησαμε δηλαδή τα κονδύλια των προπερασκευαστικών δράσεων για τον τουρισμό για όλους. Τον πρώτο χρόνο, το 2012, μελετήσαμε πρώτα απ' όλα τη ζήτηση για προσβασιμότητα στον τουρισμό και κάναμε μια σχετική οικονομική ανάλυση. Λάβαμε υπόψη μας δημογραφικά στοιχεία, πώς δηλαδή θα προχωρήσει η δημογραφική εξέλιξη, ποιες είναι οι ανάγκες του τουρίστα με ειδικέ ανάγκες και κάναμε και μια οικονομική αξιολόγηση. Μια δεύτερη μελέτη είχε να κάνει με την αξιολόγηση της προσφοράς προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την λειτουργία των ε, υπηρεσιών προσβασιμότητας στον τουρισμό στην Ευρώπη. Οπότε καταγράψαμε τις καλές πρακτικές και τις λιγότερο καλές πρακτικές. Και ασχοληθήκαμε και με την κατάρτιση, γιατί είναι ένας τομέας όπου η κατάρτιση και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν πολύ βασικά στοιχεία. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι το επαγγελματικό προφίλ που χρειάζεται κανείς και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε επίσης Ποια είναι η κατάρτιση που χρειάζεται περισσότερο για να αποκτήσει κανείς αυτό το προφίλ. Τις... Οι μελέτες ε, αυτές θα γίνουν γνωστές στα τέλη της χρονιάς, οι αρχές της επόμενης, αλλά ήδη μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία από τα αποτελέσματά τους, που πιστεύω ότι αξίζουν τον κόπο. Για την προσφορά του προσβάσιμου τουρισμού ασχοληθήκαμε ειδικά με τα άτομα με αναπηρίες. Καλές πρακτικές, marketing, πράγματα τα οποία συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται στην συνήθη προσφορά τουρισμού. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την πληροφορία, την ε, επικοινωνία και την πρόσβαση στην ενημέρωση. Mm. Λείπει δηλαδή αυτή η επαρκή ενημέρωση. Όσον αφορά την προσφορά, οι τουριστικές ε, προσβάσιμες υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως στα άτομα με σωματικές αναπηρίες και προσπαθούμε να σκεφτούμε και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των πολιτών και κυρίως μας ενδιαφέρει η ποιότητα των υπηρεσιών μας των τουριστικών. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι μεταφορές. Η έλλειψη δηλαδή μεταφορών εύκολων προς τα ελκυστικά σημεία για τον τουρισμό. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία κρίσιμα όσον αφορά την πρόσβαση. Βάσει λοιπόν αυτών των πρώτων πληροφοριών, κάναμε ένα διαγωνισμό πρόσφατα και ο οποίος έχει να κάνει με το design, με την εκτέλεση, την πρόθεση και την εμπορία ε, προσβάσιμων τουριστικών διαδρομών για να δημιουργήσουμε ένα ικανή μάζα ε, τουριστικών ε, προορισμών ώστε να φροντίσουμε συγχρόνως για τα καταλήματα, την ψυχαγωγία, shopping, ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε. Και προσπαθήσαμε, θέλουμε μάλλον, να προσπαθήσουμε να αλλάξει λιγάκι η προσέγγιση, η στάση, γιατί οι τουριστικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρίας. Η προσβασιμότητα αυτή πρέπει να ακούγεται σαν μια οικουμενική φιλοξενία όπου ο φιλοξενούμενος να είναι στην καρδιά της τουριστικής προσφοράς. Αυτά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ερωτήσει έχετε, είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι ευρωβουλευτές τώρα. Ο κύριος Δικουάνης πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους. Μας δώσατε όλοι μία σαφή προσέγγιση των ευγενών καθηκόντων και στόχων που έχετε θέσει. Η Επιτροπή και ο Πρόεδρο Σταγιάννη συνειδητοποίησαν πρόσφατα τη σημασία που έχει ο τουρισμός. Σημασία ως βασική οικονομική δραστηριότητα, έτσι, πέρα από τη σημασία που έχει ο τουρισμός για κοινωνικούς λόγους, που είναι κάτι αδιαφυσβήτητο. Παρόλο που η συνθήκη απαγορεύει την εναρμόνιση, Παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρξει συμβίωση ανάμεσα σε ένα εμπόριο, γιατί για τη χώρα μου είναι η πρώτη οικονομική δραστηριότητα. Συγχρόνως όμως καλύπτει και ανάγκες σε ένα κόσμο που η δημογραφία έχει ως έχει. Έχουμε όλο και λιγότερα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ζουν όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει με σωστό τρόπο, με δίκαιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους ενδυνάμει τουρίστες, όπως επίσης και όλα τα άτομα με αναπηρία. Το θέμα της εποχιακότητας και της προστασιμότητας λίγο πολύ είναι δύο όψεις ενός νομίσματος, γιατί ο τουρισμός είναι πολύ ανταγωνιστικός και σκληρός συχνά. Εμπόριο τι είναι, είναι να προσφέρουμε ελκυστικά πράγματα για να πετύχουμε. Και είναι θλιβερό που χώρες όπως η δικιά μου είχε μια χρονιά ιδιαίτερη γιατί, γιατί άλλες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή άλλες χώρες της ε, Αραβικής ε, Άνοιξης αποτρέπουν τον τουρισμό εξαιτία των προβλημάτων εκεί. Και γι' αυτό λοιπόν ήρθαν πάρα πολλοί τουρίστες ε, στη χώρα μου. Και είναι κρίμα που είναι αυτός ο λόγος. Τώρα, μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο τουρισμός βοηθάει την οικονομική δραστηριότητα. Χρειάζεται στήριξη για καλύτερη προσβασιμότητα υπέρ των ηλικιωμένων και μια τέτοια κοινωνική διάσταση έχει σαν αποτέλεσμα ότι η ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις που θα έκλειναν μπορούν, εφόσον υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα, η αυξημένη προσβασιμότητα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Και είναι υποχρέωση των ε, αρχών ο ιδιωτικός τομέας να βρίσκει κίνητρα ώστε να μπορεί να συμμετέχει, να έχει συμφέροντα δηλαδή, στον τουρισμό. Κάθε μέρα που περνάει, οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, λιγότερες υποχρεώσεις, οπότε εν δυνάμει είναι ένας καταπληκτικός πελάτης. Είναι καταπληκτικοί πελάτες οι ηλικιωμένοι. Δεν έχουν πια οικογενειακές υποχρεώσεις, θέλουν να ταξιδεύουν και μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν όλο και περισσότερο. Αν λοιπόν ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας φροντίσει οι τουριστικές περιοχές να είναι όλο και πιο προσβάσιμες, θα είναι η κότα με το χρυσό αυγό. Αυτό είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, η εποχικότητα δηλαδή και η προσβασιμότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους προσκεκλημένους μας και σας πρόεδρε. Ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι πλέον συμφωνούμε στο ότι ο τουρισμός δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά είναι μια ανάγκη και ένα δικαίωμα για όλους. Και συμφωνούμε επίσης ότι η δυνατότητα πρόσβασης οπουδήποτε για τον καθένα, είτε σε έναν χώρο, είτε, σε ένα, είτε στα μέσα ε, μεταφοράς, για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, και όχι μόνο τουριστικής, ε, δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μιας κοινωνίας και ενός τόπου. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι ε, μέσα στην, στην αλαζονία ε, της ε, ηλικίας μας, τους φρίγους, της υγείας μας, ξεχνάμε ότι δυνάμει είμαστε μέρος μιας επερχόμενης γενιάς ή γενεών που θα έχουν προβλήματα προσβασιμότητας, κινητικότητας και άρα μας αφορά και άμεσα τον καθένα προσωπικά και εξαιτία του δημογραφικού ε, της Ευρώπης αφορά νομίζω κάθε οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου και τον τουρισμό απόλυτα. Πρέπει να θυμίσω επίσης ότι η κάθε έκφραση του κοινωνικού τουρισμού ε, διαθέτει πολλές ευαισθησίες γιατί η ευαισθησία συνήθως δεν είναι μονοδιάστατη. Έτσι, οι εκφράσεις του κοινωνικού τουρισμού νομίζω χαρακτηρίζονται από ευαισθησίες για το περιβάλλον, ε, για ε, την κοινωνική πραγματικότητα ε, του χώρου φιλοξενίας, για ό,τι συνιστά αυτό που λέμε βιώσιμο και δίκαιο τουρισμό. Άρα θα πρέπει να είναι η έκφραση του κοινωνικού τουρισμού, κάθε έκφραση, ευπρόσδεκτη σε, σε κάθε περιοχή που, που, που εκφράζει τουριστική δραστηριότητα. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που διαρχόμαστε και που δυστυχώς έχουμε μέλλον μπροστά μας. Οι, οι, εκφράσεις του κοινωνικού τουρισμού γίνονται ή πρέπει να γίνονται όλο και περισσότερο επιθυμητές και αποδεκτές από τουριστικούς προορισμούς που μέχρι χθε έκριναν ότι δεν είχαν ανάγκη τον κοινωνικό τουρισμό γιατί απευθύνονταν κάπου αλλού. Ε, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και όλοι έχουμε βιώσει από διάφορες ιδιότητες τα προβλήματα που συναντά ε, ο κοινωνικός τουρισμός στην κάθε του έκφραση και ιδιαίτερα τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Αυτό που απαιτείται είναι η συνέργεια όλων αυτών που συνεμπλέκονται. Και εδώ υπάρχει ζήτημα και θα ήταν ευχή έργο αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε στο να υπάρξει αυτή η αποκοινού αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων και η συνεννόηση μεταξύ και των συνεμπλεκομένων της αγοράς σε όλα τα στάδια και σε όλες τις κλίμακες της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως των τοπικών κοινωνιών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κολατσέκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα τσεχικά, μια και έχουμε διερμηνία να πω ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο κλάδο στην Ευρώπη που απασχολεί 3-8% των εργαζομένων της Ευρώπης και άμεσα το 15% σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειπης πληροφόρηση, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις επαρκή πληροφόρηση, αλλά εδώ θεωρώ ότι είναι το πιο, ότι είναι το σημαντικό σημείο. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετή πληροφόρηση μέσα από ενημερωτικά δελτία, μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό που μας προκαλεί προβλήματα είτε εμένα που είμαι τρίτη φορά έχω γίνει τρεις φορές 20 χρονών ή οποιονδήποτε άλλο είναι η οποιοδηποτε αλλο ειναι η γλωσσα για παράδειγμα, της χώρας ε, προορισμού. Και αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα. Τι άλλο λείπει ε, στους ανάπηρους, για παράδειγμα, μια κοινή σήμανση των ε, οχημάτων τους. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει τελικά λυθεί και δεν υπάρχει απαραίτητα αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει να κάνει και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων με αμαξίδια. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα βαρικοίας, που έχουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά την όρασή τους. Και αυτοί θέλουν να απολαμβάνουν τον τουρισμό, τις διακοπές τους. Ίσως κάποιοι από εσά έχετε στην οικογένειά σας άτομα με αναπηρία και ξέρετε τι προβλήματα υπάρχουν. Αυτός ο ενιαίος ε, χαρακτήρας και η ενιαία διαμόρφωση της ε, αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών θα μπορούσε να ωφελήσει. Το συζητάμε για νιωστή φορά το θέμα αυτό και στα πλαίσια του αθλητισμού. Ο αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρία, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα πιστεύατε πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς τέτοιες εκδηλώσεις ε, και δυνατότητες ε, για τα άτομα αυτά. Επίσης προβλήματα παρουσιάζονται πολλές φορές στις αεροπορικές, ε, στα αεροπορικά ταξίδια. οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στα ταξίδια τους. Στην πόλη μου, ξέρετε, υπάρχουν πολλά πάρκα που δεν έχουν φράγματα, δεν έχουν φράκτες, προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν και τα άτομα με τα αναπηρικά καροτσάκια. Έχουμε χώρους ευεξίες, ε, στα σύνορα μεταξύ Τσεχίας και, ε, και Σλοβακίας. Στη Βαβαρία επίσης υπάρχουν ε, ανάλογες ε, προβλέψεις. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό λοιπόν, πρέπει να εξετάζουμε και το μη αναπτυγμένο δυναμικό. Η εποχικότητα αποτελεί λοιπόν ένα παράγοντα. Τα διάφορα είδη τουρισμού που δεν έχουν αξιοποιηθεί αποτελούν ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Χαίρομαι που τα συζητάμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Καταφέραμε εδώ να συζητήσουμε τα δύο θέματα που είναι σήμερα προς συζήτηση προσπαθώντας να επικεντρωθούμε στην εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, ώστε να είναι πιο εύκολη η λειτουργία. Όμως εγώ δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος, όχι τόσο από το περιεχόμενο, αλλά από την προσέγγιση της συζήτησης. Γιατί είμαστε επιφυλακτικοί, είμαστε διστακτικοί. Αντίθετα, θα έπρεπε να μπούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο θέμα, γιατί δεν είναι ένα θέμα που είναι ευθύνη των ε, ανθρώπων που αναλαμβάνουν ε, έκθεση για αυτό το ζήτημα. Όχι, πρέπει να υπάρχει δυναμισμός για να προχωρήσει παραπέρα το θέμα. Και έτσι να βρούμε επιπλέον επιχειρήματα. Πάντως, Ακούστηκαν διάφορα στοιχεία που για μένα πρέπει να ξεπεραστούν. Το ότι υπάρχουν μελέτες που γίνονται αυτή την εποχή για το θέμα που έχει να κάνει με την προσβασιμότητα. Είπατε ότι υπάρχει τέτοια μελέτη. Ναι, μα πριν από τρία χρόνια η Επιτροπή μας είχε τον καινούριο κανονισμό για τις στατιστικές, για τα στατιστικά δεδομένα και είχε ζητήσει να είναι δημόσια ένα σωρό στοιχεία, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν σήμερα τη βάση για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Τώρα δηλαδή επαναλαμβανόμαστε. Το θέμα δηλαδή δεν είναι να είμαστε πάντα και να παραμένουμε στο σημείο της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων, πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, επιτέλους. Γιατί οι δυνατότητες είναι τεράστιες για την οικονομία, για τους νέους, απασχόληση. Τόσοι νέοι που ψάχνουν δουλειά. Υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ μόνο σε ένα στοιχείο, έτσι ενδεικτικά. Η Ιταλική κυβέρνηση έκανε μία μελέτη σε όλη τη χώρα για τον τουρισμό και έδωσε το εξή στοιχείο. Το 2020 η Ιταλία αναπτύσσοντας διάφορα θέματα μεταξύ άλλων και αυτό έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 30 δις με 55.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερούμε, τέσσερα χρόνια έχουμε καθυστερήσει τώρα, όσο καθυστερούμε περισσότερο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα να τη χρησιμοποιήσουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ο Επίτροπος ε, Ταγιάννη έχει κάνει πολλά, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε συγχρόνως ότι μένουν πολύ περισσότερο ακόμα να γίνουν. Δύο παραδείγματα θα σας δώσω και θα τελειώσω με αυτό, Πρόεδρε. Προσβασιμότητα. Στην Ελλάδα υπάρχει σχετική εμπειρία στη Σαντορίνη που πήγα εγώ και το είδα. Και Πομπία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Πομπία κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για όσους μπορούν να περπατήσουν. Αλλά είναι μια τραγική εμπειρία για κάποιον που έχει πρόβλημα προσβασιμότητος και κάποια σωματική εμπειρία. Αυτές οι δύο εμπειρίες είναι μεν πολύ διαφορετικές, αλλά τελικά δείχνουν δύο ακραίες περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση είναι δυνατή πρόσβαση, στην άλλη δεν είναι. Και θα τελειώσω με τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισμού. Και εδώ πρέπει να οδηγηθούμε σε κάτι πιο πρακτικό. Γιατί ό,τι κάνουμε στην αρχή και στο τέλος της σεζόν μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά σημαντικά. Παλιά ο τουρισμός ήταν κάτι σνόμπ, ήταν για την ελίτ, ήταν για αυτούς που μπορούσαν να κάνουν το γύρο της Ευρώπης. Σήμερα όμως ο τουρισμός είναι κάτι θεμελιώδες για την οικονομική ανάπτυξη των ε, χωρών μας και των περιφερειών μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι, χρειάζεται ριζοσπαστική αλλαγή. Ευχαριστώ. Πριν σχολιάσουν οι εμπειρογνώμονες αυτά που είπαν οι βουλευτές, θα ήθελα και εγώ να πω ότι έχω πάει και στο Ηράκλειο και στην Πομπία, στο Ερκουλάνο δηλαδή, και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά των προβλημάτων εκεί, τα προβλήματα εκεί με αυτά που έχουμε και στις σύγχρονες πόλεις, στα κέντρα των πόλεων χωρίς καν να σκεφτούμε τους αναπήρους, η, τα καλτερίμια είναι δρόμοι που εμποδίζουν πολύ τους ανάπηρους και όποιον δεν περπατάει τέλεια. Τώρα για την εποχιακότητα. Είναι και αυτό από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες δεν θα πηγαίνουν όλοι μαζί σε τεράστιες μάζες μόνο τον Αύγουστο να επισκεφθούν χώρες. Την περασμένη εβδομάδα στο Μάντσεστερ ας πούμε ήταν το κέντρο γεμάτο παιδιά, αυτή την εβδομάδα γεμάτο συνταξιούχους γιατί τα παιδιά πήγαν όλα στο σχολείο. Επομένως το θέμα δεν είναι να ελέγξουμε τις τουριστικές ροές ακριβώς, αλλά να οργανωθούν καλύτερα οι τουριστικοί οργανισμοί. Γιατί όταν υπάρχει τέτοια συρροή αυξάνονται και οι τιμές. Δηλαδή γίνονται πιο ακριβές οι διακοπές με παιδιά και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τέτοιες διακοπές παίρνουν τα παιδιά τους διακοπές βγάζοντάς τα από το σχολείο. Αυτό είναι δύσκολο και πρέπει εδώ και οι τουριστικοί πράκτορες κάτι να κάνουν, να μοιράσουν κάπως τις προσφορές ώστε να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές όχι μόνο τον Αύγουστο. Είναι σαν την έξοδο που σημειώνεται στο Παρίσι την πρώτη εβδομάδα τον Αύγουστο. Πρέπει να το δουν οι ψυχολόγοι αυτό. ιδίω στα διόδια του Κλερμό Φεράν να πάνε ψυχολόγοι και να δούνε ότι υπάρχουν εκεί άνθρωποι που περιμένουν 20 και 24 ώρες για να περάσουν τα διόδια. Μήπως θέλουν οι εμπειρογνώμονες να κάνουν κανένα σχόλιο. Βιτάλε, κύριε Βιτάλε, θέλετε να πείτε τίποτα. Για δύο λεπτά όμως μόνο. Καλά. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την τάση να δημιουργήσουμε πρότυπα για την αγορά αυτή. Ο στόχος είναι ο κάθε τουρίστας ατομικά και οι ανάγκες του. Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά μόνο τους αναπήρους, αλλά και δημιουργεί, δεν αφορά μόνο τους αναπήρους, αλλά δημιουργεί και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αν υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα, τότε ικανοποιείται περισσότερο και ο τουρίστας και η αγορά εργασίας. Υπάρχει ένα λογισμικό που συλλέγει στοιχεία για ικανοποίηση των κριτηρίων που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αλλά πάντως δεν θέλουμε στερεότυπα και ακίνητα πρότυπα, αλλά την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των τουριστών. Πρέπει να λυθούν προβλήματα που αφορούν και δημόσιους και ιδιωτικούς τρόπους μεταφοράς. Ας πούμε, αν μπορεί κανείς να ανεβεί στο τρένο εύκολα με αναπηρική καρέκλα ή στο αεροπλάνο. Άμα θέλουμε να βελτιωθεί η εποχιακότητα, τότε πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα πάρα πολλών ανθρώπων και συχνά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μην επενδύσουν σε διαφορετικούς τρόπους οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Θα ήθελα επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην πληροφόρηση των επιχειρηματιών των ίδιων για να γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξουν και αυτές οι νέες αγορές. Να συμφωνήσω με τον προηγούμενο μελητή. Αυτά που ισχύουν για τους ανάπηρους συχνά ισχύουν και για τους ηλικιωμένους. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα πρέπει να φοράμε μία ετικέτα στο κεφάλι ή πού να τη φοράμε την ετικέτα. Ότι έχουμε την τάδε ή δίνα αναπηρία. Όταν γνωρίζουμε ότι οδεύουμε προς μία κοινωνία η οποία θα έχει πιο πολλούς ηλικιωμένους, δεν θα είναι ατομικό ζήτημα, θα είναι το ζήτημα, ξέρετε, όλη η κοινωνία που γυράσκει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι στο, για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούμε ως κοινωνία και οι αρχές θα πρέπει να προετοιμαστούν. Άρα όλο και πιο πολλές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και να αποχωριστούμε τα σημερινά στερεότυπα. Είτε είσαι ηλικιωμένος που τρως τα λεφτά της κοινωνίας για να φας τα λεφτά σε τουριστικούς προορισμούς ή είσαι κάποιος που εξαρτάσαι από κάποιον άλλον, είσαι εξαρτώμενο άτομο. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θα μπορούσα να κάνω κατάχρηση της θέσης μου. Έγινα 60 χρονών τον Φεβρουάριο. Έγινα... Ε, ε, με... Βγήκα στη σύνταξη. 5 Φεβρουαρίου ήμουν μεσήλικας και μετά 6 Φεβρουαρίου έγινα ηλικιωμένο. Για πείτε μας κι εσείς, σε ό,τι αφορά την εποχικότητα, είναι σημαντικό να μην οδηγούμε, εξαναγκάζουμε τον τουρίστα να ταξιδεύει κάποιες συγκεκριμένες εποχές. Για παράδειγμα, αυτό μας απασχόλησε και εμάς, γιατί έχουμε σήμερα 55.000 προσφορές στην πλατφόρμα μας Όλες αυτές οι προσφορές έχουν να κάνουν σε περίοδους χαμηλής σεζόν. Γιατί όλο αυτό φυσικά αποτελεί πηγή ε, εσόδων και οικονομικής ισορροπίας, αλλά και οι ταξιδιώτες σε κάποιες περιπτώσεις ε, επιθυμούν να ταξιδέψουν κάποιες συγκεκριμένες περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική ενημέρωση, αν θέλετε, να δώσουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Είδαμε στην αγορά των ε, ηλικιωμένων, αλλά και με τα άτομα με αναπηρία. Αυτοί οι ίδιοι από μόνοι τους προτιμούν τις πιο νεκρές εποχές, γιατί είναι πιο άνετο το ταξίδι. Είναι πιο χαλαρωτικό, δεν υπάρχει τόσο άγχος, δεν υπάρχει περιοθώριο σύγχυσης, αλλά συχνά παρατηρείται ένα πρόβλημα παράλληλων υπηρεσιών. Είναι κλειστά τα μουσεία, δεν παρέχονται συγκεκριμένε υπηρεσίε και έτσι έχουν κάποια προβλήματα όταν τελικά ταξιδεύουν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη σε περιοχές χαμηλής ε, επισκεψιμότητας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πρότυπο και κανόνες για το πώς θα ορίζεται η προσβασιμότητα. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα θέμα ενιαίας κατανόησης, αν θέλετε, του όρου. Και σημειώνω εκ νέου σε ό,τι αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, ότι κάποιες χώρες έχουν ε, μία ετικέτα, αν θέλετε. Κάθε χώρα έχει μία ετικέτα. Όταν ταξιδεύω όμως με χώρα, με ε, ομάδα με ανάπηρους, ε, στη Φλάνδρα για παράδειγμα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω απαραίτητα πάντα αυτές τις ετικέτες, γιατί δεν είναι κοινέ παντού. Θα πρέπει να είναι κοινέ όμως, για να ξέρει ο ταξιδιώτης τι να περιμένει. Ο κύριος Μπορκίνη. Mm, Θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρατήρηση, αλλά χωρίς να σας καθυστερώ, είμαστε σε έναν τομέα που έχει πολύ σημασία η, προ... η ζήτηση και η προσφορά. Γι' αυτό και θα είμαι προσεκτικός. Όταν λέμε να παρατείνουμε την τουριστική σεζόν, ξεκινάμε από την ανάλυση μιας ζήτησης που υπάρχει ήδη. Ξεκινάμε δηλαδή από την αρχή που λέει ότι υπάρχει η προσφορά αλλά η ζήτηση είναι περιορισμένη σε ένα-δύο μήνες. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν η ζήτηση των ηλικιωμένων που είναι περισσότερο διαθέσιμη. Φυσικά υπάρχουν και τα συνέδρια που βοηθούν τον τουρισμό. Υπάρχουν οι νέοι που μετακινούνται, σπουδάζουν αλλού. Υπάρχει ο αθλητισμός, υπάρχουν δηλαδή αθλητικές δραστηριότητες ή πρωταθλήματα που λαμβάνουν χώρα εκτός σεζόν. Ας βασιστούμε λοιπόν περισσότερο στη ζήτηση. Αν θέλουμε έναν τουρισμό μεγάλης κλίμακας, ας ξεκινήσουμε από τις ανάγκες κινητικότητας, ας ξεκινήσουμε από αυτό που ενδιαφέρει τους κατοίκους, οι οποίοι θέλουν να μπορούν να έχουν υπηρεσίες ποιότητας και πρόσβαση παντού. το πρόγραμμα που ξεκίνησε είναι πολύ ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα Καλυψό καθόρισε τέσσερις τυπολογίες. Αλλά κανονικά υπάρχουν και άλλες. Όλοι μιλούν για τους νέους, για τους ηλικιωμένους, για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μετά βάζουμε και τους ανάπηρους. Όχι. Βέβαια, είναι ένας τρόπος για να αρχίσει κανείς να δουλεύει, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ένα άτομο με αναπηρίες που έχει προβλήματα θα τα παντού ως πολίτης. Για να έχουμε λοιπόν τουρισμό ποιότητας, πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε όλους τους δυνατούς χώρους για να γίνουν πιο ορατά τα προσόντα μιας περιοχής. Ο κύριος Σανταντέρ. Ναι, γιατί στην προσβασιμότητα θέλω να αναφερθώ κι εγώ. Συγγνώμη αν υπάρχει ήδη νομοθεσία, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για όλες τις χώρες μέλη όσον αφορά τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Μιλήσατε πριν για διαφορετικές ταμπέλες. Ναι, το να είναι κανεί σε ένα ξενοδοχείο σε μια χώρα είναι εντελώ διαφορετικό από το να είναι σε ένα ξενοδοχείο ακόμα και αν έχει τον ίδιο αριθμό αστεριών, α πούμε, σε μια άλλη χώρα. Εγώ προσωπικά είμαι από τον ιδιωτικό τομέα. Θα σας δώσω στοιχεία, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, θα σας τα αφήσω. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας. Είναι από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας του 2012 τα στοιχεία αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ένα εκατομμύριο άτομα έχουν κάποια ε, αναπηρία, το 1 τρίτο του πληθυσμού, πάλι από την ίδια οργάνωση, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτό σημαίνει 15% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβει την οικονομική σημασία που μπορεί να έχει αυτή η κατηγορία ατόμων για τον τουρισμό και για την οικονομία γενικότερα. Θα λέγω ότι είναι ένας κλάδος που μπορεί να ηγηθεί της οικονομίας μας, εφόσον πρόκειται για τόσο κόσμο. Πρέπει να επευθεθούμε λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα για ένα θέμα που δεν μπορεί να λυθεί από το δημόσιο τομέα, να ζητηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και να μπορεί να έχει κέρδος από εκεί. Πρόεδρος, ναι, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Μιλάμε για την προσβασιμότητα και σωστά για τα άτομα με αναπηρίες. Προβλήματα κινητικότητας. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου για την προσβασιμότητα οικογενειών με μικρά παιδιά και ως παππούς δεν κάνει μηνών είναι τον κόνη μου. Είναι θέμα αυτό, ειλικρινά σας το λέω. Μερικές φορές για να οδηγήσετε το καροτσάκι και να κυκλοφορήσετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να δούμε και την προσβασιμότητα των οικογενειών με μικρά παιδιά. Και το άλλο που θέλω να θίξω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε Welcome to Europe, καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Ωραία, αναφερθήκατε και στις θεωρήσεις. Είναι πρόβλημα. Ο έλεγχος διαβατηρίων είναι πρόβλημα. Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη μας λέτε, ναι και το πρώτο πράγμα που σας λέει η Ευρώπη, όταν πάτε τουλάχιστον στον Ηνωμένο Βασίλειο, είναι τι, 35 λεφτά περιμένετε για έλεγχο διαβατηρίων. Δεν έχετε καν μπει στη χώρα. Ε. Και το δεύτερο που θέλω να πω για το Welcome to Europe, τι εννοείται ακριβώς Welcome ε, τι, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη. Η υπόλοιπη Ευρώπη, η πραγματική Ευρώπη, αυτή που βρίσκεται στο πρόγραμμά σας. Παρακαλώ κύριε Τουντίνη, για πείτε μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω στο θέμα της προσβασιμότητας. Στις μελέτες που κάναμε, ορίσαμε όντως ως προσβάσιμο τουρισμό ε, το προσβάσιμο του τον τουρισμό σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με προσωρινά σωματικά προβλήματα και οικογένειες με μικρά παιδιά. Περιλαμβάνονται λοιπόν. Δεν θέλαμε να εξαιρέσουμε οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα. Θέλαμε να έχουμε περιμετρική κάλυψη, αν θέλετε, των αναγκών των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Ναι, όχι. Για άλλο θέμα μιλάμε. Η καμπάνια μας, η ενημερωτική, θέλει να περάσει το μήνυμα ότι η Ευρώπη αποτελεί μία ομάδα πολλών διαφορετικών προορισμών. Προωθούμε λοιπόν την Ευρώπη στο σύνολό της. Πρόκειται για μία εκστρατεία που περιλαμβάνει και άλλες δράσεις χάρη στο Κοινοβούλιο, όπως η πρωτοβουλία είδαμε για παράδειγμα για την προώθηση μη παραδοσιακών προορισμών. Συγχρηματοποιούνται λοιπόν από τις ομάδες μας project που έχουν να κάνουν με παραδοσιακούς, ε, δεν θα βρείτε στο πακίτο μας μάλλον, παραδοσιακούς προορισμούς, γιατί είναι αρκετά ισχυροί από μόνοι τους. Δεν μας χρειάζονται οι προορισμοί που μας χρειάζονται είναι οι μικροί προορισμοί. Και νομίζω ότι τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο μικρών προορισμών. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ήταν ένα από τα πράγματα που περιλήφθησαν στο Eden, στο πρόγραμμα αυτό σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική για τις θεωρήσεις. Ξέρουμε ότι ο έλεγχος διαβατηρίων μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι τελείως εκτός της σφαίρας ελέγχου μας. Εργαζόμαστε για τον νέο κώδικα για τις θεωρήσεις. Θα έχει ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το τέλη του έτους. Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμοστούν κατά πάσα πιθανότητα το 2015 για τις ε, θεωρήσεις, αλλά θέλουμε να ενημερώσουμε και τα κρατη για το πώς θα πρέπει να εφαρμόσουν τις ήδη υφιστάμενες ε, προδιαγραφές. Υπάρχουν ε, νομικά έντυπα για τα αεροδρόμια, για τα προξενία. Αυτό λοιπόν μπορεί να ευαισθητοποιήσει, αλλά τελικά εξαρτάται από τα κρατη να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Υπάρχουν οι διατάξεις, υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές, ξέρουμε ότι είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνει ένας επισκέπτης από την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις τεράστιες ουρές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κάρλο, θα ήθελες να συνοψίσεις. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, γιατί Υπάρχουν μερικές διαφορές απόψεων εδώ που δείχνει, πράγμα που δείχνει πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα, αλλά και επίσης ότι είχαμε δίκιο που το συζητούμε. Παραδείγματο χάρη, υπήρξαν διαφορές ως προς το θέμα των προτύπων. Ακούσαμε για βέλτιστες, λέει, πρακτικές που ξεπέρνουν το θέμα των απλών προτύπων και αφορούν τη μεταχείριση των ανθρώπων σε ατομική βάση. Άλλοι επιμένουν σε ανάλυση πιο δομική. Το πόσοι και ποιοι τουρίστες δηλαδή προτιμούν το α ή το β ξενοδοχείο ή προορισμό. Και άλλοι πάλι ζητούν μία ολόκληρη εναρμόνιση. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα θέμα που θα συνεχίσει να συζητιέται και θα χρειαστεί περισσότερη εμβάθυνση. Ταυτόχρονα δεν ξέρω αν ήταν, είχε υποθεί επίτηδες, αλλά ακούστηκε και η ιδέα ότι οι ανάπηροι, οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι ίσως οι καταλληλότεροι για να ξεπεράσουν το θέμα του εποχιακού περιορισμού. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση τελικά, αλλά υπάρχει και το θέμα του τι, μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την αποεποχιακότητα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι ή ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα αποκλειστικά για τον Αύγουστο. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στο μέλλον σε όλα αυτά. Και το τελευταίο θέμα που πρόσεξα, είναι κάτι που το έχουμε ξαναπεί αλλά θα πρέπει ακόμη να το ξαναδούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αρκετά χρήματα για μετεκπαίδευση και πληροφόρηση και έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θέλουμε να περιοριζόμαστε μόνο στις πληροφορίες και τα συμφέροντα των τουριστικών οργανισμών, των ξενοδοχείων, δηλαδή των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τομέα. αλλά ότι θέλουμε να τους οθήσουμε και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τουριστών. Αυτό σημαίνει βέβαια και διαφορετικού είδους πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα, χωριστό. Τέλος, τελευταίο σχόλιο αφού είμαστε Επιτροπή Μεταφορών δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πρόβλημα που ανέφεραν όλοι την προσβασιμότητα στις μεταφορές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για προσβασιμότητα ορισμένων κατηγοριών τουριστών, αυτό αφορά καταρχήν τη μεταφορά τους. Και εδώ πρέπει να το ξαναδούμε και σας ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε και τους συναδέλφους αλλά ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες σήμερα που ήρθαν να μας κάνουν αυτήν την πολύ χρήσιμη συζήτηση. Καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερους συναδέλφους αλλά τις πέμπτες το απόγευμα έτσι γίνεται. Πάντως είναι σημαντικό τμήμα των ενδιαφερόντων μας στην Επιτροπή Μεταφορών αυτό που συζητήσαμε σήμερα και όπως είπε και ο κύριος Κόλιτσεκ στην Ευρωπαϊκή Οικονομία αφορά και την Ευρωπαϊκή Οικονομία στο σύνολό της και την ανεργία και τις θέσεις απασχόλησης. Θα οργανώσουμε και άλλες στρογγυλές τράπεζες. Ελπίζω να συνεχίσει να προσέρχεται η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ όλους για όσα είπατε σήμερα. Για τους βουλευτές σας υπενθυμίζω την επόμενη μας συνεδρίαση Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 3. Και εδώ ευχαριστώ και το προσωπικό και τους διερμηνείς και κηρύσσετε το πέρα της συνεδρίασης.